Uh, Είστε έτοιμοι λοιπόν. Έχουμε μόνο ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά πριν περάσουμε στην ψηφοφορία θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνουμε μία δοκιμαστική. Για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Σας καλώ λοιπόν να βάλετε τις κάρτες σας. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μία δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. I close Πέρα της δοκιμαστικής. Όχι ακόμα. Λοιπόν, θέλω να ξαναδοκιμάσουμε. Δεν πρόλαβαν όλοι οι συνάδελφοι. Παρακαλώ πολύ και πάλι μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Σας παρακαλώ όλους να προσπαθήσουν να ψηφίσουν. Είστε όλοι εντάξει. Μπορούμε να περιμένουμε ένα λεπτό. Έχω ξεχάσει ε, την κάρτα μου στις ψηφοφορίες της ΙΜΚΟ. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτάκι για να έρθει. Αν είναι ένα λεπτό, κανένα πρόβλημα. Διαφορετικά ε, θα σας λαμβάνουμε υπόψη δεδομένου ότι δεν έχετε την κάρτα. Για να δούμε λοιπόν. Sorry, let's vote uh, draft uh, Λοιπόν, για το σχέδιο του ψηφίσματος για την αναθεώρηση ε, των κατευθυντηρίων γραμμών για ε, τις ε, ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη. Ήταν προφορική τροπολογία της Ήτρε. Πέρασε το θέμα από το Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, υπέρ, κατά ή αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία. Είστε εντάξει, συνάδελφε. Ωραία. Πέρα τη ψηφοφορία. 70, 55, 15 κατά και τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν το ψήφισμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξη που είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προπολογισμό του 2021, τμήμα τρίτο. Σας υπενθυμίζω πως οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές είναι το πρώτο ψήφισμα το οποίο εγκρίνει στα πλαίσια της διαδικασίας προπολογισμού του Κοινοβούλιο έτσι ώστε να παρουσιαστούν οι προσδοκίες του Κοινοβουλίου για το προπολογισμό του επόμενου έτους. Το ψήφισμα θα εγκριθεί τον Απρίλιο στην Ολομέλεια και ε, στέλνουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ε, το ψηφίσουμε. 45 λεπτά θα αφιερώσουμε στην συζήτηση αυτή και θέλω να το θεωρήσετε μια ευκαιρία, ε, συνάδελφοι, ε, τουλάχιστον εσείς που είστε τμήμα των διαπραγματεύσεων για το δημοσιονομικό, για τις πολιτικές δημοσιονομικές πρόπτικες. Θέλω λοιπόν να μου κάνετε κάποια σχόλια, να μας πείτε τι συμβαίνει στις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τι συμβαίνει εκεί γενικότερα και παρακαλώ οι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο να ε, σηκώσουν το χέρι τους. Ε, και μάλιστα αντί να σηκώσουν το χέρι σας προτείνω να σηκώσετε ε, το καρτελάκι σας τοποθετήστε το κάθετα έτσι ώστε να σας δει η γραμματεία και να σας σημειώσει. Okay. By saying this... Ωραία λοιπόν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και θα πω δύο λόγια ως εισηγητής για το θέμα αυτό. Αγαπητοί και συνάδελφοι, αγαπητοί σκιώδεις, αγαπητοί εισηγητέ για τα διάφορα προγράμματα, δεδομένου ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα συμφωνία για το ΠΔΠ, οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό αυτό θα πρέπει να απηχούν τη γενικότερη στάση μας για το θέμα των ΠΔΠ και για τα προγράμματα που έχουμε στην εντολή της ΙΤΡΕ, δηλαδή το νέο πρόγραμμα την νέα αγορά, το Horizon, το InvestEU κτλ. Για τις κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν για τον προπολογισμό του 2021, να σας πω πως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταθεί στεναρά, να υπερασπιστεί ε, το ε, στόχο που έχει, ε, έτσι ώστε ε, να ε, έχουμε την πρικοδότηση που ζητούμε γιατί το Συμβούλιο προτείνει πολύ χαμηλότερα ποσά για το ε, πρώτο τίτλο να σας πω πως για την ψηφιακή ε, μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα, την βιομηχανική, τη μετάβαση στα ενεργειακά ε, σε συμφωνία με τα όσα είπαμε στο Παρίσι, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα κονδυλία, κυρίω για την ψηφιακή μετάβαση, έτσι ώστε να μην εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Οποιαδήποτε μείωση κάτω από αυτό που προτείνει στο πρόγραμμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Connecting Europe θα πρέπει να απορριφθούν κατά τη δική μου γνώμη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές και για εμάς και για την Ευρώπη. Αποτελούν αναπόσπαστο κρίσιμο τμήμα της οικονομίας και η μετάβαση από το πρόγραμμα COSME στο νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και για το ΕΦΣΥ ε, θα πρέπει να γίνει με τα κατάλληλα εργαλεία μέσω του Invest EU. Εμείς εδώ και χρόνια δίνουμε τη μάχη για να έχουμε ένα δίκαιο ταμείο μετάβασης και θα συνεχίσουμε και στα πλαίσια αυτά ε, περιμένουμε ε, την ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε την σημαντική συμβολή των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εφαρμοστούν οι πολιτικές αυτές που χρειάζονται λοιπόν χρηματοδότηση και η Ανίσα και η GSA και η BEREC που χρειάζονται ε, και ε, το απαραίτητο προσωπικό και τον απαραίτητο προϋπολογισμό. Τέλος, όλοι αναγνωρίζουμε ε, ε, πόσο σημαντικό είναι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης. Είδαμε ε, τα ποσά που προτείνει ο Πρόεδρος, κύριος Μισελ, και κατά τη γνώμη μου, και σίγουρα αυτό το συμμερίζονται αρκετοί συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αρκετές άλλες προεδρίες επιτροπών, δεν επαρκούν. Το Horizon Europe είναι κάτω από τη φιλανδική πρόταση του Δεκεμβρίου. Ε, το facility για την, ενέργεια, για την ενέργεια και για τα ψηφιακά είναι πολύ χαμηλότερα από τις προτάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για το Digital Europe ακόμα χαμηλότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λίγο καλύτερα από τη Φιλανδική, ε, για το διάστημα λίγο καλύτερα από τη Φιλανδική πρόταση που ήταν 30% αν θυμάμαι καλά κάτω, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από τα όσο θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Άμυνας είμαστε αρκετά υψηλότερα, αλλά η κινητικότητα των στρατιωτικών έχει μειωθεί, το οποίο σημαίνει ότι εξουδετερώνεται το οποιοδήποτε πλεονέκτημα τη αύξηση. Και έχουμε και παραπάνω περικοπέ στι υπηρεσίε που έχουμε σε, όλα, ε, σε όλους τους τίτλους ε, του προπολογισμού. Είναι πολύ διαφορετική λοιπόν η πρόταση από αυτή, από την πρόταση που εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν τη συζήτηση και τροποποιήσεων και κατά τη γνώμη μου θα θέσει σε κίνδυνο τη δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τι νέε προκλήσει και τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε μελλοντικά. Σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις, δύο λεπτά ο καθένας και μετά θα έχουμε και τον κατάλογο έτσι ώστε να ακούσουμε τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους οι οποίοι κάτι θέλουν να πούν. Δίνω το λόγο κατευθείαν στους σοσιαλιστές. Η κυρία Γκάλβες Μουνιός παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τα βασικά θέματα που θέσατε κύριε Πρόεδρε και πρέπει να σας πω πως ανησυχώ και θα το εκφράσω για την καθυστέρηση, για τη συμφωνία ε, για, τα, για τις ΠΔΠ και αυτό θα έχει αρνητικές και συγκεκριμένες συνέπειες. Για παράδειγμα, προγράμματα έρευνας. Η καθυστέρηση αυτή σημαίνει απόλυτα 5.000 ε, θέσεων ερευνητών το μήνα που θα επηρεάσει και πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Όπως είπατε και εσείς κύριε Μπουσόη, δεν μπορούμε να δεχτούμε μία πρόταση για το Horizon Europe, η οποία να είναι κάτω από την ήδη πολύ χαμηλή πρόταση που έχει καταθέσει η Φιλανδική Προεδρία. Στηρίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, την, τον τίτλο 1 που είναι η ενιαία αγορά ε, και τα ψηφιακά για να τονίσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους κλάδους αυτούς για να αντιμετωπίσουμε επίγουσες ε, περιστάσεις όπως για παράδειγμα η επιχειρηματικού ουδετερότητα μέχρι το 2050, όπως επίσης και μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά βρίσκονται στον κόμβο του Ευρωπαϊκού Green Deal και ευθυγραμμίζονται με τα όσα έχουμε αναλάβει στα πλήση της Συμφωνίας των Παρισίων ως μακροπρόθεσμους στόχους. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για ένα φιλόδοξο σχέδιο προπολογισμού, κάτι το οποίο στηρίζεται από την Προεδρία των Τεσσάρων Ομάδων ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το πρόγραμμα για την ψηφιακή αγορά, έτσι ώστε να έχει τα όπλα που θα επιτρέψουν με κυριαρχία να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ψηφιακή πρόκληση. Έρευνα και ε, ανάπτυξη. Εδώ έχουμε μεγάλο κενό επενδυτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γύρω στα 110 δις, τόσο έχει ε, ε, υπολογιστεί κατ' και αυτό θα πρέπει να το καλύψουμε. Και για το πρόγραμμα για το διάστημα και εκεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι επενδύσεις θα βρεθούν για να πετύχουμε τους στόχους του Green Deal. Ίσως χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο να προωθήσουμε ε, νέους επιπλέον ίδιους πόρους. Για παράδειγμα, είτε ένα φόρο επί των αεροπορικών ε, ε, μετακινήσεων είτε ε, υπέρ του κλίματος είτε επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για να καταφέρουμε να υπερασπιστούμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε για τα επόμενα έτη. Διαφορετικά διακινδυνεύουμε. Θα χάσουμε το τρένο του μέλλοντος. Και αυτό θα κάνει όλο και πιο δυσαρεστημένους με την Ευρωπαϊκή Ένωση τους ε, πολίτες μας και θα αποστραφούν όλο και περισσότερο την ίδια τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκάλβες ε, Μινιός. Η κυρία Βαλερή Χάιρ εκ μέρους της Renew. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Είναι καλή η πρότασή σας και για τη Renew να σας υπενθυμίσω τρία σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα μας. Και γι' αυτό ε, θα τα πω πριν τα υποβάλω ως τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα, σας τα υπενθύμησαν, θα πρέπει ε, για τους ίδιους πόρους να μετασχηματίζουμε το πώς βρίσκονται αυτοί. Προσωπικά να σας πω πως είμαι και κομμάτι των διαπραγματεύσεων και για τους ίδιους πόρους συνεισηγήτρια, οπότε για τους ίδιους πόρους το έχουμε πει δεν θα ψηφίσουμε ε, τις πι δέλτα πι ε, αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί χρειάζεται να κάνουμε πρόοδο και να βρούμε καινούριου ίδιου πόρου. Δεύτερον, μικρομεσαίε επιχειρήσει και στήριξη αυτών θα πρέπει και αυτές να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό για να αναπτυχθούν. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το υπογραμμίσατε και εσείς, η ανάγκη να υπερασπιστούμε προγράμματα όπως ψηφιακή Ευρώπη έτσι ώστε να μπορέσουμε τις κομβικές επενδύσεις στην τεχνολογία του αύριο να τις κλειδώσουμε τη μία πάνω στην άλλη και να εξασφαλίσουμε και την κύβερνο ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ ο προπολογισμό του 2021 διαφέρει αρκετά από τον προηγούμενο. Γι' αυτό και εμεί οι πράσινοι σκεφτόμαστε ότι ε, θα πρέπει και η άποψη μα να είναι ισχυρότερη από τα προηγούμενα χρόνια. Λόγω του ΠΔΠ, οι διαπραγματεύσει, όπω όπως είπε και η Σασά, συμμετέχω και εγώ στι διαπραγματεύσει και όπω βλέπουμε τώρα υπάρχουν πολλέ προτάσει επιτάπητο. εκτό όμως από την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου στο να φτάσουμε στους κοινούς μας στόχους, όπως τους στόχους για το κλίμα, δεν το, την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 ή νωρίτερα ή και την δαπάνη του 3% των κονδυλίων για ερευνητικά προγράμματα. Βλέπουμε όμως περικοπές στα προγράμματα που αφορούν την Επιτροπή μας. Πιστεύουμε ότι ε, τα δικά μας, ε, ίσως επίσης να πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα για τα αγροτικά προγράμματα και τα πρόγραμματα σύνοχης και θέλουμε εξυγχρονισμό του προπολογισμού και του ΠΔΠ και των περικοπών του προγράμματος ορίζοντας. Ε, έχουμε ακούσει από τους άλλους συναδέλφους, είναι προβληματικά, αλλά και άλλα προγράμματα, αν δούμε τους αριθμούς, μας απογοητεύουν, περιλαμβάνουν σημαντικά θέματα, υπάρχουν περικοπές και εκεί πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς, να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην ομάδα των διαπραγματεύσεων και των ευρωβουλευτών που ε, δουλεύουν σε αυτό και γι' αυτό ο ρόλος της Επιτροπής μας είναι σημαντικός όχι για τους αριθμούς αλλά και για την ποιότητα. Και θα πρέπει να διεξάγουμε κάποια συζήτηση για το πρασίνισμα του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και έχουμε και μια συζήτηση για την ε, εξάλληψη των ορυκτών καυσίμων θα ε, είχαμε κάποιες ε, αποφάσεις. Ελπίζουμε όμως να προχωρήσουμε και σε αυτό το μέτωπο και να έχουμε ένα πιο ε, δυνατό προπολογισμό για το 2021. Ευχαριστώ. Έχουμε τρεις συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Ξεκινάω φυσικά με τον κύριο Νίκα Συντονισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με τα κονδύλια για τον ορίζοντα Ευρώπης, θα ήθελα και εγώ να πω ότι το ποσό δεν είναι επαρκές. Αν στον ορίζοντα του 2020 αν είχε, υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότητας ε, ενός έργου στα 10, ταυτόχρονα με αυτή την ε, δραματική περικοπή των κονδυλίων για τον ορίζοντα Ευρώπης ε, και τα προγράμματα τα ερευνητικά θα έχουν δυσκολίες δεν είναι σαφείς οι προτεραιότητες, γιατί αν ταυτόχρονα βλέπουμε ότι θα έχουμε επενδύσεις απαραίτητες για ε, για το υδρογόνο ως νέα μορφή ενέργειας, ε, ε, επενδύσεις στις ορευτές και άλλα για την Πράσινη Συμφωνία και ταυτόχρονα έχουμε περικοπές στις πηγές χρηματοδότησης, ε, που θα πρέπει να περιλάβουν αυτές τις νέες και τόμες ε, τεχνολογίες. Νομίζω εδώ είναι μια μεγάλη παγίδα, γι' αυτό ε, θα ήθελα να απορρίψουμε αυτές τις προτάσεις στο, στο θέμα των, της έρευνας. Και δεν είναι επίσης σαφές πώς θα λειτουργήσει Έχουμε ένα ταμείο που το ζητήσαμε, το Ταμείο Μετάβασης και το κονδύλι που έχει κατανεμηθεί σε αυτό το... είναι συζητήσιμο γιατί είναι μικρό. Αλλά από αυτό το κονδύλι που ε, δόθηκε ε, στις, ε, για την βοήθεια στις επιχειρήσεις για να περάσουν στο phase out των ορυκτών καυσίμων και έχουν εντοπιστεί κάποιες περιφέρειες στην Ευρώπη που υπάρχουν ενεργοβόρες βιομηχανίες και έχουμε φτάσει σε ένα θέμα που ισχύει και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ε, εμφανίζεται σε όλα όσα ζητάμε και αυτά τα προγράμματα για την εξάλληψη του άνθρακα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν γι' αυτό αντί να έχουμε στόχο το 2030 για την εξάλληψη του... Θα, θα φτάσουμε στο 2050. Αυτό θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί. Θα πρέπει να ξέρουμε όλοι τι μας περιμένει. Και θα πρέπει να ξέρω κι εγώ ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη ε, όταν ε, προτείνονται τέτοιες προτάσεις. Ε, εάν δεν θα γίνει το Green Deal, τότε να μας το πούνε ξεκάθαρα και στα ράτα. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε ξεκάθαρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλλετε. Είμαι σίγουρος ότι θα μεταδώσετε αυτά τα μηνύματα. Loud and clear, όπως λέμε στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Νίκα. Ε, το σημειώνω και στηρίζω την προσέγγισή σας. Ο κύριος Τάσνοντεύσκη έχει το λόγο τώρα. Του με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Ε, Děkuji, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να σας ευχαριστήσω και να σας πω πως εκτιμώ ιδιαίτερα την ποιότητα της έκθεσής σας κύριε Κρασνιδέση και να υπογραμμίσω τα εξής δύο. Γιατί αναφερθήκατε και εσείς σε αυτά. Καταρχήν να σας πω πως στηρίζουμε, στηρίζουμε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα. Είναι μια υπηρεσία η οποία θα ε, υποκαταστήσει, θα αντικαταστήσει μάλλον τις δύο προηγούμενες τις υπηρεσίες GNR και GNS και είναι οι δύο υπηρεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνε για τα προγράμματα Κοπέρνικους και Γκαλιλαίου στην Ευρώπη. Να σας πω όμως πως ε, δεν έχουμε, και αυτό με δυσαρεστεί, την αύξηση οικονομικών πόρων και ανθρώπινων πόρων για αυτή την υπηρεσία. Ξέρετε πως έχουμε πάρα πολλά χρόνια που συζητάμε για τα θέματα αυτά, για το Γαλιλαίο και η Επιτροπή μας πολύ συχνά έχει ζητήσει οι ανθρώπινοι πόροι και οι οικονομικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι να αυξηθούν και αυτό δεν μοιάζει να έχει επηρεάσει καθόλου την κατάσταση και δεν βλέπουμε καμία τέτοιου είδους αύξηση. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσω για την ε, υπηρεσία Μπερέκ και εκεί τα καθήκοντα όλο και αυξάνονται, η τεχνολογία τρέχει και για μια φορά ακόμα θα πρέπει και εδώ να ζητήσουμε μια αύξηση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων διαφορετικά η ΠΕΡΕΚ δεν θα μπορεί να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της. Στηρίζω την ε, ε, γνωμοδότησή σας, την έκθεσή σας και οι τροπολογίε μου θα είναι σχετικές με αυτά τα οποία μόλις τώρα σχολίασα. Thank you so much, Mr. Uh, next speaker is uh, Mr. Gair, Ο κύριος Γκάλ, από τους Σοσιαλιστές, παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά θέματα τα οποία έπτυξαν οι συνάδελφοι και συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις για το πολιτέ σε δημοσιονομικό πλαίσιο, θα ήθελα να επισημάνω ένα θέμα στους συναδέλφους, ότι πριν από 7 χρόνια αυτή τη χρονική στιγμή, δηλαδή μέσα Φεβρουαρίου, ε, ήμασταν έτοιμοι με τις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Και μέχρι όμως να εφαρμοστούν όλα τεχνικά μέχρι τα Εθνικά Κοινοβούλια να ακυρώσουν ε, τον κανονισμό περί ιδίων πόρων, μέχρι να συνταχθούν ε, λειτουργικά προγράμματα. Ε, πέρασε η χρονιά χωρίς κατ' ουσίαν να εκταμιευτούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν για μας ότι ενδομεταξύ είμαστε στα μέσα Φεβρουαρίου και από ό,τι προβλέπετε την Πέμπτη δεν θα υπάρξει συμφωνία. Άρα δηλαδή αν τα συγκρίνουμε με το τι έγινε το 2013 σε αντίθεση με ό,τι είχαμε συμφωνήσει έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Και όλα αυτά σημαίνουν αν δούμε και τα προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή κατά την τεχνική εφαρμογή των προγραμμάτων. Αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας, ε, φοβάμαι ότι το 2020-2021 θα είναι μια χαμένη χρονιά και αυτό για μας ε, στην Ήτρε σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ λιγότερα κονδύλια από ό,τι επιθυμούσαμε στην ε, πολιτική, κοινή πολιτική έρευνας. Φοβάμαι λοιπόν ότι στην Ευρώπη δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μα τέτοιου είδου πολυτέλειε, αν δούμε τι γίνεται στην τεχνολογία και στην έρευνα. Εγώ λοιπόν στηρίζω τους συναδέλφου ε, όσον αφορά τα στοιχεία και τους αριθμούς του Πουδουπού, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να βιαστούμε λιγάκι για να μην χαθεί η χρονιά 2021. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γκρουντλέρ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμμερίζομαι αυτά που είπατε. Είναι σημαντικό. Στο θέμα του διαστήματος, όπως είπε και ο συνάδελφος, όπως και εσείς είχατε πει, ότι είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι το Κοινοβούλιο ζητούσε 16,9 δις για το ΠΔΠ και είμαστε πολύ μακριά από το στόχο και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν για τον προπολογισμό του 2021 ήδη να έχουμε τουλάχιστον την συντήρηση, ε, να διατηρήσουμε κάποιους ε, στόχους που είχαμε ήδη θέσει. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Θα πρέπει να έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με τα μέσα ε, για τους διάφορους οργανισμούς. Το GSA φυσικά το έχετε θυμίσει. Ε, ο οργανισμός GSA είναι ευρωπαϊκός οργανισμός που δεν έχει τα μέσα να λειτουργήσει. Ε, όμως έχει σημαντική αποστολή που δεν μπορεί να την εκπληρώσει. Υπάρχει η GSA αλλά και οι άλλοι παίκτες, οι άλλοι οργανισμοί που είναι απαραίτητοι για να τρέξει το πρόγραμμα, που είναι σημαντικό για να έχουμε το φιλόδοξο αυτό σχέδιο που έχουμε για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Χάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεσή σα. Αυτή η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την βιομηχανία στην Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίσει ότι έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία, ιδιαίτερα στην απανθρακοποίηση της ε, ε, βιομηχανία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αν θέλουμε να έχει απόδοση η Πράσινη Συμφωνία. Όπως ε, ξέρουμε είναι βαριές οι βιομηχανίε που δεν έχουν ακόμη βρει τι λύσει για την απαλλαγή από τις ανθρακουχείς εκπομπές μέχρι το 2000, ε, το 2050 είναι ο απόλυτος στόχος. Ε, θα πρέπει όμως να κινηθούμε πιο γρήγορα όπως γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης. Εάν η έρευνα και η οτομία ε, ε, ενισχυθούν, τότε θα γίνει πρόοδος ταχύτατα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η έρευνα, ιδιαίτερα ορίζοντας έχουν επαρκή χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίση να διασφαλίσουμε ότι και τα κονδύλια που πάνε στον ορίζοντα ε, συμμετέχουν και στην Πράσινη Συμφωνία, έτσι ώστε να μην δαπανώνται κονδύλια σε τεχνολογίες που τελικά να μην ε, ε, μας βοηθήσουν για τους στόχους βιοπικιλότητάς μας. Σας ευχαριστώ κυρία Πάουλους. Τέλος, ο κύριος Χάιζελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχέδιο της έκθεσης. Πολύ καλή έκθεση και ισορροπημένη. Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι λείπουν κάποια κονδύλια για πολύ σημαντικά προγράμματα έρευνας για το πρόγραμμα Horizon. Από την άλλη πλευρά θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρεστε στη σημασία της εισαγωγής ε, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό αν θέλουμε να έχουμε ε, μια επιτυχημένη μετάβαση και να μην ζημιωθούν οι ευάλωτοι πολίτες. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι χρειαζόμαστε όχι μόνο ε, σταθερή χρηματοδότηση, αλλά και το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης θα πρέπει να προέρχεται από ε, φρέσκο χρήμα, γιατί αλλιώ, όχι δηλαδή από το Ταμείο Συνοχής, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο συνοχή ε, θα ε, ευεργετούνται στο μέλλον λιγότερο. Ω εκ τούτου, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε πραγματικά νέα κεφάλαια, φρέσκο χρήμα, Προς το παρόν, με πάση περιπτώσει, είμαι ικανοποιημένος και ε, θέλω να πιστεύω ότι θα επιτύχουμε μια περισσότερο ισορροπημένη συμφωνία που να αφορά στα κράτη-μέλη. Πρόεδρος, αν δεν υπάρχουν ε, άλλες ε, παρεμβάσεις, επιτρέψτε μου εγώ να πω λίγα λόγια κλείνοντας αυτή τη συζήτηση για τον ε, προϋπολογισμό να ευχαριστώ την εισηγήτρια, τις σκιώδη εισηγήτρια, ε, Γκουγιές Μουνό, ε, Εράσμους Άντερσεν, ε, να τους ευχαριστήσω για τις προτάσεις που κατέθεσαν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε αποφασιστικότητα υπερασπιζόμενη το όραμά μας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους ίδιους πόρους και κάτι που ανέφεραν η κυρία Χάιερ και ο κύριος Άντερσεν αναφέρθηκαν στην ψηφιακή Ευρώπη. Η ψηφιακή Ευρώπη ε, πρέπει να παραμείνει πολύ σημαντική. Αν περικόψουμε κονδύλια από την ψηφιακή Ευρώπη ε, θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ανταγωνιστικό ε, περιβάλλον να είμαστε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο. Ε, όσον αφορά την έρευνα, το πρόγραμμα Horizon ε, θα πρέπει να χρηματοδοτείται σωστά. Αυτά που προτείνονται σήμερα είναι απαράδεκτα. Και βεβαίω το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση που ανέφεραν η κύριοι Νίκα και Χάιζελ, αυτό το ταμείο είναι πολύ σημαντικό ε, για εκείνε τι ε, περιφέρειε που αντιμετωπίζουν προβλήματα και βεβαίως χωρίς την υποστήριξη των ευρωπαϊκών κοντιλίων για νέες τεχνολογίες, νέες επενδύσεις και νέες θέσεις απασχόλησης ε, είναι σχεδόν αδύνατον ε, για αυτή την, αυτές τις περιοχές να εφαρμόσουν την Πράσινη Συμφωνία. Αυτό όμως ε, είναι ένα στρατηγικός στόχος. Όλοι συμφωνούν από αυτού. Επ Οι δύο επόμενοι συνάδελφοι ε, συμφώνησαν για τα ειδικά προγράμματα για τα εξωτερικά γραφεία. Ε, επίσης υπάρχει το πρόγραμμα για το διάστημα το οποίο υποχρηματοδοτείται και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να αγωνιστούμε επίση πολύ σκληρά. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σα καλέσω να καταθέσετε τροπολογίες. Ε, είμαι σίγουρο ότι τελικά θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο έγγραφο και θα έχουμε και πολύ καλύτερη θέση αν επανεπιβεβαιώσουμε τις προτεραιότητές μας και το όραμά μας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ε, Αυτά όλα για τα επόμενα 7 χρόνια. Βέβαια, η πρώτη χρονιά είναι το 2021 και θα πρέπει να ξεκινήσουμε ευθύ εξ αρχή ε, προ τη σωστή κατεύθυνση. Σα ευχαριστούμε πολύ για τι ε, παρεμβάσει σα ε, και θα ήθελα παρακαλώ να μην ξεχάσετε ότι η καταληκτική προθεσμία είναι η 19η Φεβρουαρίου στις 12 η ώρα, καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών. Ο κύριος Πεκαρίνενεν. Έχω να υποβάλω άλλη μια ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κονδύλια για την Πράσινη Συμφωνία, κυρίως ε, στις περιοχές όπου υπάρχει άνθρακας, για να μπορεί να γίνει μετάβαση. Είναι όμως επίσης ε, σημαντικό να υπάρχουν κονδύλια και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, για τον εξυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ε, για να μην υπάρξει μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Οποτεδήποτε επενδύουμε νέα σύγχρονη τεχνολογία στη βιομηχανία μας, ε, τότε δεν υπάρχει και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Είναι σημαντικές οι ε, περιοχές άνθρακα, αλλά είναι επίσης σημαντικό να ε, μειωθούν οι εκπομπές αερίων. Συμφωνώ απόλυτα και πιστεύω πως και εδώ θα πρέπει να βρούμε κάποιες εναλλακτικές, καθαρές, νέες τεχνολογίες. Θα λάβουμε βεβαίως υπόψη και τη δική σας συνεισφορά. Μην ξεχαστείτε, μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου μπορείτε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας και με αυτά κλείνουμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό για να περάσουμε στα γρήγορα στο σημείο 10 Πάμε καλά χρονικά. Έχουμε 45 λεπτά για την έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος ISA 2. Κυρία Γκέρτρουτ Ινκεστάτ, σας καλωσορίζω. Είχα τη χαρά να σας συναντήσω το Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της σημερινής συνάντησης της Ήτρε. Κυρία Ινκεστάτ είναι η Γενική Διευθύντρια για την πληροφορική από τη Γενική Διεύθυνση ε, Digit και Έχουμε τώρα τη δεύτερη φάση του προγράμματος ε, για τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια έκθεση αξιολόγησης 23 Δεκεμβρίου του 2019 και η συνέχεια για το πρόγραμμα αυτό θα δοθεί από το πρόγραμμα ε, Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ευρώπη, η οποία επίσης ανήκει στη καθήκοντα της Ήτρε. Θα μας παρουσιάσετε λοιπόν ε, τα σχέδια για την ψηφιοποίηση της δημόσιας δίκης στην Ευρώπη στο μέλλον και τα σχέδια γενικότερα της υπηρεσίας για το μέλλον. 45 λεπτά στη διάθεσή μας και παρακαλώ όσοι συνάδελφοι θέλετε να πάρετε το λόγο ε, να μας βοηθήσετε να καταγράψουμε το ενδιαφέρον συμμετοχής με τον νέο τρόπο που είναι πιο αποτελεσματικός και πιο εύκολος, με τις καρτελίτσες σας δηλαδή κάθετα. Και η κυρία Ίγκεστα τώρα έχει το λόγο, σας δίνω 10 λεπτά να κάνετε μια αρχική παρουσίαση και μετά θα ακούσουμε τους συντονιστές ή τους αντικαταστάτες, τους αναπληρωτές, τον κύριο Ζωρίνιο, άλλα μέλη. Δύο λεπτά ο καθένας και μετά Είπαμε δύο λεπτά οι συντονιστέ και ο κύριο Ζωρίνια και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από ένα λεπτό και στο τέλο θα ξαναδώσουμε το λόγο για τουλάχιστον πέντε λεπτά στην κυρία Γενική Διευθύντρια για να αποκριθεί με λεπτομέρειε τα όσα θα ρωτήσετε. Κυρία θα σα δίνω το λόγο. Thank you very much, dear... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε Μπουσόη. Αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποδέχεστε εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη χαρά και για μένα και για την ομάδα μου, γιατί είμαστε αρκετοί εδώ, να είμαστε εδώ ενώπιον ε, της Εκλεκτής Επιτροπής αυτής, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι η Επιτροπή Ήτρε που παρακολούθησε και στήριξε το πρόγραμμα διαλειτουργικότητας 2016-2020. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω τον κύριο Κάρλο Ζωρίνιο και τους σκιώδεις εισηγητέ για τη στήριξη στο πρόγραμμα ΙΣΑ 2. Σήμερα είναι χαρά μου να σας παρουσιάσω τα κυριότερα σημεία της αξιολόγησης του προγράμματος ΙΣΑ 2, της παραμονές της οριστικοποίησης του. Επίσης, με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για το μελλοντικό όραμα για την ψηφιοποίηση των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Διοικήσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ε, έντιμα Το πρόγραμμα ίσα στο τετράγωνο στηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που καθιστούν δυνατό για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στην Ευρώπη να επωφεληθούν από διαλειτουργικές, διασυνοριακές και διατομεακές δημόσιες υπηρεσίες. Έχει τους ακόλουθους στόχους. Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητε επιτάχυσης της διαλειτουργικότητας ε, ε, συντονίζονται καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασυνοριακά, να αναπτύξει και να λειτουργήσει λύσεις για τις δημόσιες διοικήσει με βάση του τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, επίσης να θεσπίσει τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία για την τόνωση της διαλειτουργικότητας σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα ένα αναθεωρημένο ευρωπαϊκό δίκτυο πλαίσιο διαλειτουργικότητας, μια αναθεωρημένη ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας, το ΕΙΡΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Αναφορά στη Διαλειτουργικότητα, τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων το TPE... Ε, σε προτινόμενη ε, νομοθεσία ευρωενωσιακή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, νέκρινε την έκθεση στα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος ΙΣΑ 2 στις 23 Σεπτεμβρίου του 2019. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 109 ερωτηθέντα ενδιαφερόμενα μέρη, εκτεταμένη δευτερογενή έρευνα και πραγματογνωμοσύνες, η ενδιάμεση αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι οι επιδόσει του προγράμματος ίσα στο τετράγωνο είναι καλές ω όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Ε, συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνεχτικότητα, προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία, χρησιμότητα, βιοψημότητα. Οι στόχοι που ακολουθεί το ίσα στο τράγωνο είναι ε, σημαντικοί και εναρμονίζονται με τους ε, στόχους. Ε, το Η υλοποίηση του προγράμματος προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα με ισχυρή εσωτερική συνοχή ανάμεσα στις διάφορες δράσεις του ίσας τετράγων. Η ε, ικανοποίηση των χρηστών με τις λύσεις, η... για παράδειγμα το EU Survey, Join Up, Leos, που στηρίζει την σύνταξη νομοθεσίας. Αυτά είναι θετικά, η ικανοποίηση είναι θετική. Το πρόγραμμα ενίσχυσε τις σχέσεις με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα άλλα προγράμματα ε, κυριότερα είναι η ευκολία ΣΕΦ, η διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη ΣΕΦ, ορίζοντα 2020 και το πρόγραμμα στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι ε, που επαναχρησιμοποιούν ή προωθούν ε, τις λύσεις ίσα στο τετράγωνο. Επίσης, ίσα στο τετράγωνο αλληλεπιδρά με πρωτοβουλίες όπως είναι το Single Digital Gateway, την ε, ψηφιακή στρατηγική της ενιαίας αγοράς, το σχέδιο δράσης e-government, την διακήρυξη του Ταλίν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ε, και ιδιαίτερα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν για την προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η απουσία του θα διακύβευε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα και να τονώσει τον εξυγχρονισμό του δημοσίου τομέα στην Ευρώπη μέσω ΤΑΦΠΕ. Βέβαια, υπάρχουν και τομεί που χρήζουν βελτίωση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσωπική μα περισσότερο στο να ευαισθητοποιήσουμε πέραν από τι εθνικέ διοικήσει προ τι περιφερειακέ και τι τοπικέ διοικήσει. Δουλεύουμε με στοχευμένε δραστηριότητε για να, τονώσουμε, να τονίσουμε με τα πλέον εκτήματα επαναχρησιμοποίηση των λύσεων ιδιαλειτουργικότητα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ίσα στο τετράγωνο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Πρωτοβουλία Ακαδημίας Διαλειτουργικότητας που ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο του 2019 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λόιβεν. Στοχεύει να ενθαρρύνει δημόσιες διοικήσεις, τον ακαδημαϊκό κόσμο και ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές. Θα ήθελα επίσης να προτείνω αυτή την πρωτοβουλία και να σας καλέσω να ε, συμμετέχετε ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία. Τι ακολουθεί τώρα. Είμαστε πεπισμένοι ότι όταν τελειώσει το ίσα στον τράγωνο θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να το χρησιμοποιήσουμε ως μια νέα βάση για να κτίσουμε και να διαμορφώσουμε ε, πλήρως ψηφιοποιημένες δημόσιες διοικήσεις σε όλη την Ένωση ως απαραίτητο θεμέλιο για, να, ε, για μια ψηφιακή Ευρώπη. Η τεχνολογική πρόοδος μας δίνει τα μέσα να πετύχουμε αυτό για τους πολίτες. Ε, χάρη στην τεχνολογία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων και των πιο αποκλεισμένων. Άρα το ψηφιακό έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίζει τις δημόσιες διοίκησεις και να τους δίνει τη δυνατότητα να παραδίδουν τις υπηρεσίες τους σε ένα σταθερό, αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο. Αυτή είναι μια ε, τεράστια ευκαιρία ε, για τον ευρωπαϊκό δημοσιοτομέα και είναι η ευκαιρία που μας δίνεται αυτή τη στιγμή. Και από αυτή την άποψη ο Επίτροπος Χάν έλαβε την αποστολή να ε, πρωτοστατήσει με το στόχο της ε, ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών δημοσίων δικήσεων, ξεκινώντας με την ίδια την Κομισιόν. Η Κομισιόν θα ηγηθεί με το παράδειγμά της. Ο δικός μας ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μοναδική ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό της ψηφιοποίησης, να δημιουργήσουμε καινοτόμες λύσεις για ε, μια πιο αξιόπιστη, αποτελεσματική, αποδοτική και διαφανή και ασφαλή Κομισιόν. Θα συγκεντρωθούμε σε δράσεις που θα επιταχύνουν αυτό το μετασχηματισμό έτσι ώστε η Κομισιόν να γίνει ένας ψηφιακός οργανισμός πανέτοιμο για τις προκλήσεις τη ψηφιακή της ψηφιακής εποχής. Ε, ψηφιακή στρατηγική που υιοθετήθηκε πριν από 18 μήνες περίπου και οι συνέργειες και αποτελεσματικότητες, αυτή η πρωτοβουλία, έχουν ε, ξεκινήσει ε, αυτό τον οδικό χάρτη για να κτίσουμε ένα ψηφιακό οικοσύστημα μέχρι το 2022 με χαρακτηριστικά όπως την ιδιωτικότητα με σχεδιασμό, διαλειτουργικότητα με σχεδιασμό κλπ. Θέλουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική ψηφιακή ατζέντα ε, προς ε, την υπηρεσία και τη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών δημοσίων διοικήσεων. Τα περισσότερα συστήματα στην Κομισιόν συσχετίζουν τον θεσμό μα με τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η διαλειτουργικότητα θεωρείται ω προτεραιότητα σε τομείς όπω είναι οι μεταφορέ, η έλεγχη των σύρνόρων, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η υγεία. Η εναρμόνιση των ψηφιακών υποδομών και των προτύπων, η υιοθέτηση και η επαναχρησιμοποίηση των λύσεων και των μοντέλων διαλειτουργικότητας είναι ε, βασική ε, κινητήριος δύναμη για την ψηφιοποίηση, για να δημιουργήσουμε διασυνοριακές ψηφιακές υπηρεσίες. Άρα είναι σημαντικό να αντανακλώνται αυτές οι προτεραιότητες στο επόμενο πι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογούμε και να προωθούμε τις προδιαγραφές και τα πρότυπά μας. Και στόχος μας είναι να επιταχύνουμε και να βελτιώσουμε ψηφοποίηση των δημοσίων διοικήσεων σε όλη την Ένωση. Αυτό ισχύει για την Κομισιόν, για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και για τις δημόσιες διοικήσει ε, της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα. Προτεραιότητα μας θα πρέπει να είναι να απλουστεύσουμε περίπλοκες διαδικασίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες καθημερινά, για παράδειγμα, τις διασυνοριακές φορολογικές δηλώσεις, ηλεκτρονικές ταυτότητες, την εγγραφή τους σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος. Η ψηφιακή δημόσια διοίκηση θα επιτρέψει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη να υποφεληθούν από τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες ανεξαρτήτως του από πού προέρχονται και πού που ζουν ή που δουλεύουν. Οι, ε, καλά, οι ψηφιακές δημόσιες διοικήσεις που λειτουργούν καλά θα ε, έχουν ε, μειωμένη Γραφειοκρατία επίσης. Για αυτούς τους λόγους ε, ερχόμαστε εδώ για να ζητήσουμε τη συνεργασία σας, γιατί θεωρούμε ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου είναι σημαντικός. Θα ήθελα κλείνοντα να πω ότι θέλουμε να δουλέψουμε μαζί σα, να, σας, να ακούσουμε τι προτάσει σα, να μάθουμε από την εμπειρία σα στι δικέ σα εκλογικέ περιφέρειες και να σα καλέσουμε να δουλέψετε μαζί μα για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γενική Διευθύντρια, για την ε, παρουσίασή σα. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για όλα αυτά που έχετε επιτύχει. Ε, και τώρα έχουν το λόγο οι συντονιστέ, οι οι αναπληρωτέ των συντονιστών και μετά θα λάβει το λόγο ο κύριο Ζωρίνιο. Και υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο εκ μέρου του ΕΛΚ, η κυρία Καρβάλιο, επειδή δεν είναι παρόντε όλοι οι συντονιστέ από τι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε, ε, να μου πείτε ε, ποιο ε, θέλει να λάβει το λόγο αντικαθιστώντας συντονιστή, αλλιώς θα περάσω στα μέλη. Εγώ, αν θέλετε, ε, θα μιλήσω ο συντονιστής. Η κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Γενική Διευθύντρια. Έχω τέσσερις ε, συστάσεις. Ε, πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για τη δουλειά σας και έχω τέσσερις συστάσεις οι οποίες βασίζονται στην ε, εμπειρία μας, στις εκλογικές μας περιφέρειες, στην εμπειρία μας και ως πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό Κατά τη διάρκεια της ε, ψηφιοποίησης της ε, δημόσιας διοίκησης να ε, θεωρήσουμε ότι είναι μια ευκαιρία να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες και να μην προκύψουν επιπρόσθετα πράγματα σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Δηλαδή να μην έχουμε επικάλυψη διαδικασιών και βεβαίως αυτό πολλές φορές εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Η δεύτερη πρότασή μου είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα ε, όσο πιο φιλικό προς το χρήστη Δεν αναφέρομαι μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και στους πολίτες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, μερικές φορές ε, δεν συμβαίνει αυτό εξακολουθούμε να έχουμε ε, περίπλοκες πλατφόρμες ε, που καλούμεθα να χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Άρα δηλαδή ε, εδώ έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτή είναι η δεύτερη πρότασή μου. Η τρίτη αφορά στο θέμα των δεξιοτήτων. Χρειαζόμαστε βασικές δεξιότητες ε, και πάλι ε, για τους πολίτες, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γενικότερα για όλους. Αλλά χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους εμπειρογνώμονες εμπειρογνώμονες για την ψηφιοποίηση, την πληροφορική και την επικοινωνία εμπειρογνώμονες λοιπόν. Και το τέταρτο που θέλω να πω είναι κάτι που με ανησυχεί περισσότερο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε γυράσκοντα πληθυσμό ε, και αυτό ε, δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα. Γιατί ο γυράσκον ε, πληθυσμός κυρίως εντοπίζει σε χώρες που προχάνε πάρα πολύ με την ψηφιοποίηση και η τρίτη ηλικία οι ηλικιωμένοι ε, αισθάνονται κατά κάποιον τρόπο ότι απειλούνται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας. Εγώ αυτές τις προτάσεις είχα να καταθέσω. Ευχαριστούμε κυρία Καρβάλιο, ο κύριος Ζωρίνιο και είναι ε, επίσης εισηγητής. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την έκθεση, να ευχαριστήσω την κυρία Γενική Διευθύντρια και την ομάδα της. Εγώ ήμουνα εισηγητής και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο συνεργαστήκαμε και στο πρόγραμμα ΙΖΑ επιφέραμε φιλόδοξα σχέδια στη χρηματοδότηση, στην απλούστευση των διαδικασιών. Ε, κυρίως όμως όσον αφορά στα αποτελέσματα, αυτά αποτελέσματα για τον πολίτη και για τις επιχειρήσεις. Και σήμερα λοιπόν, σε αυτή την ενδιάμεση έκθεση, διαπιστώνουμε ότι βελτιώνεται η συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές διοικήσεις, στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, στους συνοριακούς ελέγχους. Όλα αυτά δείχνουν ότι ε, τα φιλόδοξα προγράμματά μας κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν. Είμαι λοιπόν ικανοποιημένος και θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα ε, της Γενικής Διευθύντριας ε, για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά αποτελέσματα. Αυτά τα καλά αποτελέσματα οδηγούν στο ότι πρέπει να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες στο μέλλον. Οι επόμενες ε, φάσεις του προγράμματος ΙΖΑ το πρόγραμμα τρέχει μέχρι το 2022 και μέχρι τότε καλούμεθα να αποδείξουμε την προστιθέμενη αξία. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γύρουμε μία γέφυρα ε, προς την ψηφιακή Ευρώπη. Ε, αυτό κατά τη Φιλανδική Προεδρία είχε χαθεί, αλλά κάπως επανήλθε και η Κροατική Προεδρία το έχει συμπεριλάβει πάση περιπτώσει έχουμε ε, μια ισχυρή ψηφιακή Ευρώπη. Εγώ είμαι σκιώδη ηγητή τη πολιτική μου ομάδα επί του θέματο. Νομίζω ότι η μετάβαση πρέπει να είναι απόλυτα σαφή δεν νομίζω ότι ε, είναι καλό να χρησιμοποιεί κανείς εικόνες, γιατί αυτό δημιουργεί προβλήματα στους διερμηνείς, αλλά αυτή είναι μία απλή εικόνα. Με την τεχνολογική αλλαγή δεν χρειαζόμαστε μόνο ε, αυτοκινητοδρόμους όπου να τρέχουν τα αυτοκίνητα, αλλά χρειαζόμαστε και χώρους στάθμευσης. Ε, χώρους στάθμευσης όπου να μπορεί κανείς να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε πληροφορίες για τις επιχειρήσεις για να μπορούν και αυτές να αναζητήσουν λύσεις. Το θέμα δεν είναι μόνο το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Υπάρχουν πέντε επίπεδα ε, να υπάρχει δυνατότητα λογιστική και επίσης ε, να υπάρχουν δεξιότητες και διαλειτουργικότητα. Όλα αυτά τα χρειαζόμαστε ε, για να λειτουργεί το πρόγραμμα και οι διαδικασίες και αυτές είναι και οι βάσεις ε, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες. Τώρα την αλλαγή πώς ε, θα την επιτύχετε όταν θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Δώστε μου όλα δύο δευτερόλεπτα πρόεδρε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αυτή την διάσταση πώς μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε στη συνεργασία με τους εταίρους μας γιατί πρόκειται για ένα γεωπολιτικό καθήκον. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά και δεν θα ήθελα να ταπανίσω περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζωρίνιο. Ο κύριος Νίνης το παρακαλώ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που κάνατε. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό και θα ήθελα να μιλήσω πιο πολύ για τις ε, συγκεκριμένες ανησυχίες που διακατέχουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Βεβαίως η ψηφιοποίηση και η διαλειτουργικότητα και η δημόσια διοίκηση ουσιαστικά φέρνουν σε μια ελευθερία κίνηση, σε μια καλύτερη αγορά εργασία στην δυνατότητα παροχής δημοσίων υπηρεσιών σε ε, αλλοδαπό κράτος Θέλω να μου πείτε λοιπόν εσείς, τα ε, κράτη-μέλη είναι το ίδιο δραστήρια, έχουμε διαφορές στην ε, προσπάθεια που κάνουν και να σας πω πως εγώ έχω ζήσει και στη Φιλανδία και στη Σουηδία και επειδή έχω και τις δύο επικοότητες είδα πως ε, εμείς έχουμε διασυνοριακά θέματα και ενώ 50 χρόνια το συζητάμε όταν χρειάστηκε να βγάλω σουηδικό διαβατήριο για τα παιδιά μου. Είχα φιλανδικό διαβατήριο μεν και δεν ήταν αρκετό για να εξηγήσω ότι είμαι ο πατέρα των παιδιών μου όταν του έβγαλα σουηδικό διαβατήριο. Χρειάστηκε να βγω στον δρόμο να μαζέψω δύο Σουηδού για μάρτυρε και να πάμε να αποδείξουμε ότι είμαι και Σουηδό. Αυτό είναι λίγο παράλογο. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε αυτέ τι ευρωπαϊκέ οδηγίε πώ τι εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη και τι γίνεται και με τα θέματα ε, τη μετανάστευση για να μην έχουμε συνοριακά προβλήματα. Δηλαδή, είναι απλή ψηφιοποίηση, απλή διαλειτουργικότητα να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε αυτά να τα ομαλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Γενική Διευθύντρια. Ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστούμε που μας ε, παρουσιάσετε το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε για τις πρωτοβουλίες σας μα μας εντυπωσίασαν. Και να ρωτήσω πρώτα απ' όλα, μήπως έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς ακριβώς μπορούν να υποφεληθούν οι πολίτες από το πρόγραμμα ΙΖΑ. Γιατί για μας αυτό είναι σημαντικό. Θέλουμε στις εκλογικές μας περιφέρειες ε, να μπορούμε να δείξουμε το πώς ωφελούνται οι πολίτες ε, από την Ευρώπη. Και η δεύτερη παρατήρησή μου είναι μια μεγάλη θερμή παράκληση προς εσάς. Στη δική μου την πατρίδα, τη Γερμανία, ε, ε, υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός γιατί πρέπει κανείς να πάρει ένα πιστοποιητικό Α1 λέγεται έτσι ώστε ε, όταν κάποιος εργαζόμενος μεταβεί σε ένα άλλο κράτος μέλος να είναι κοινωνικά ασφαλισμένος. Αυτό καλό είναι για να αντιμετωπίζεται η λαθρεργασία, η μαύρη εργασία αλλά ξέρετε αυτό είναι μια τεράστια γραφειοκρατία να πρέπει κανείς να αποκτήσει αυτό το πιστοποιητικό. να λοιπόν μια ιδανική περίπτωση ε, για να έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα clearing το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους πολίτες και τους ελεκτές. Ε, αυτό θα βοηθήσει στο να αντιμετωπιστεί η μαύρη εργασία, να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω πραγματικά θερμά να σας παρακαλέσω ε, να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα σήμερα. Μπορεί κανείς μέσα σε δευτερόλεπτα να αποκτήσει το clearing ηλεκτρονικό ε, αυτό το α 1 αυτό το πιστοποιητικό, να το μπορεί κανείς να το αποκτά ηλεκτρονικά. Και αυτό θα ήταν καταπληκτικό, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό θα διευκόλυνε ε, τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ε, ελεγκτές και αυτοί θα βλέπουν ότι είναι πολύ εύκολο να εκμεταλλευτούν την κοινή αγορά. Κυρία Πατρίτσια Τόγια, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά μου αρέσει πολύ αυτό το πρόγραμμα. Συγχαρητήρια και βεβαίω ε, ε, πράγματι αυτό παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον και για μα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το είπαν και άλλοι ε, συνάδελφοι, ότι εμείς ε, βεβαίως και είμαστε βουλευτές, αλλά είμαστε και απλοί πολίτες ε, και εμείς ε, καλούμεθα να έρθουμε σε επαφή με τη δημόσια διοίκηση. Και αν ψηφιοποιηθεί η δημόσια διοίκηση θα απλουστευτεί η ζωή του πολίτη. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο όμως πρέπει να σας πω ότι δημιουργεί και πολύ μεγάλη επιφύλαξη, τουλάχιστον στη δική μου τη χώρα. υπάρχουν πειράματα που δεν έχουν αποδώσει, άρα δηλαδή είναι ένα θέμα, θα έλεγα, αρκετά περίπλοκο. εσείς βέβαια αποδείξατε ότι μπορούν να γίνουν πράγματα, υπάρχουν θετικές πρωτοβουλίες ε, και εγώ απλά ε, θέλω να πω ότι να εκμεταλλευτείτε συγκεκριμένα ε, παραδείγματα. Γιατί αν υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, μόνο έτσι μπορεί κανείς να πείσει άλλες δημόσιες διοικήσεις. Ξέρετε, πρέπει οι εθνικές, περιφερειακές, τοπικές διοικήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η διαλειτουργικότητα είναι είναι εκ των, ουκ, κάνευ. Ε, δεν είναι ότι καλούμεθα να επανακαλύψουμε τον τροχό. Ε, γι' αυτό λοιπόν, ε, κύριε Πρόεδρε, ε, να είμαστε λίγο πιο επιτακτικοί απέναντι στις δημόσιες διοικήσεις. Νομίζω αυτό μπορούμε να το κάνουμε, γιατί αν προκύπτει κάτι καλό, γιατί να μην το χρησιμοποιούν όλοι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συγκεκριμένοι και να προσπαθούμε να διαδώσουμε τις καλές πρακτικές. Άλλος κανείς, εάν όχι να πω και εγώ δύο λόγια και να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι για την επιτυχία ε, των όσων έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Αυτή τη στιγμή έχετε εφαρμόσει πολύ ενδιαφέροντα project και είναι ξεκάθαρο πως η ψηφιοποίηση επηρεάζει όλους και χαίρομαι που θα συνεχίσετε και στο μέλλον. Είμαι βέβαιος δε πως έχετε και την πολιτική στήριξη ε, του, συνόλου των επιτρόπων και σίγουρα και την πολιτική στήριξη της Επιτροπής Ήτρε, γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Να σας ρωτήσω δε το εξής. Σε ποιο βαθμό μπορείτε εσείς να παρέμβετε στο διάλογο που γίνεται με τα κράτη-μέλη. Καταρχήν γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ του επίπεδου ψηφιοποίησης δημόσιας δημόσιας μεταξύ κρατών μελών. Και δεν είναι μόνο γεωγραφικό, γιατί μπορεί κανείς στην ίδια γεωγραφική ζώνη να βρει κανείς κάποιο πιο ε, ψηφιακά φιλοδόξο κράτος μέλος και νομίζω ότι ακόμα και στα νέα κράτη-μέλη συμβαίνει αυτό. Αυτές οι διαφορές θα πρέπει να ξεπεραστούν και πρέπει να παροτρύνουμε τις χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμα ε, πετύχει την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης ε, να το κάνουν. Funds from cohesion policy and not only which uh, could be used for uh, digitalization. Να σας πω λοιπόν <laughs> πως στη δική μου χώρα, τη Ρουμανία, τα προγράμματα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ρώτησα α, τον, α, να, τότε που ήμουν πρόεδρος λοιπόν εγώ που του Εθνικού Συστήματος ε, Υγείας ε, ε, και κοινωνικών ασφαλίσεων ε, να εφαρμόσουμε την ηλεκτρονική κάρτα υγεία. Το ίδιο έκανε και ο κύριο Νίκα, ο οποίο ήταν και υπουργό υγεία στη χώρα μα και το κάναμε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Πείτε μου λοιπόν στι επόμενε πι δελτα από τα ταμεία συνοχή και από άλλα εργαλεία πόσα κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν στα κράτη-μέλη την ε, ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και ευχαριστώ που με ακούσατε με τόση προσοχή. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Έχουμε πετύχει πολλά με το πρόγραμμα Ίσα στο τεράγωνο. Το κάναμε με την συμμετοχή πολλών κρατών μελών. Έχουμε ένα δίκτυο, λέω, υπάρχει ένα, ένα δίκτυο ε, υπό την ηγεσία κάθε κράτους μέλους. Αυτό είναι ένα σημαντικό δίκτυο που έχουμε για να συζητάμε με τα κράτη-μέλη πώς να μοιράζονται εμπειρίε, πώς να κάνουν ανταλλαγέ για τα θετικά που ισχύουν στη μία και στην άλλη χώρα. Είναι μια ευκαιρία που έχουμε δύο φορές το χρόνο. Επίσης έχουμε την Επιτροπή που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΙΣΑ 2 ε, που ε, καθοδηγεί ε, και τι πρέπει να γίνει από πλευρά των Ευρωπαίων πολίτων, πολιτών, τι χρειάζονται, ποια είναι τα κενά, ποιε είναι οι λύσεις που πρέπει να εξετάσουμε, ποια είναι τα πρότυπα που πρέπει να αναπτυχθούν. Αυτά είναι τα σημεία επαφή. Αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι Έχουμε τη βάση, τα θεμέλια, το πλαίσιο, τι κατευθυντέ γραμμέ και τι συστάσει, πολύ δυνατέ συστάσει. Έχουμε μεγάλη συνεργασία. Τώρα πώ θα πάμε στο επόμενο στάδιο, να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Αυτό θέλουμε να δούμε πώ επιταχύνουμε για να φτάνουμε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα για του πολίτε. Αυτό που σκεφτήκαμε και μελετήσαμε με του συμμετέχοντε από τα κράτη-μέλη είναι να έχουμε αυτό που είπε ο κύριο Σορίνι. Αυτός ο χώρο στάθμευση, ε, εκεί όπου έχουμε όλα αυτά τα πράγματα από του θεσμού, από τα προγράμματα, όχι μόνο το πρόγραμμα ΙΣΑ, αλλά και τα άλλα προγράμματα. Έχουμε λύσεις από την διευκόλυνση Connecting Europe, το πρόγραμμα ΙΣΑ, συνεργασία με τα άλλα προγράμματα, για να βρούμε τις συνέργειε και θα πρέπει να τις σταθμεύσουμε κάπου με ασφάλεια, όπου να έχει καθένας πρόσβαση, αλλά και τις λύσεις από τα κράτη-μέλη. Πολλά κράτη-μέλη έχουν πάρα πολύ καλέ λύσει που μπορούν να τι μοιραστούν με άλλα κράτη-μέλη. Ένα παράδειγμα που θα αναφέρω, σε μια από τις πρώτες συναντήσεις που κάναμε με τις κυβερνήσεις, είπαν ότι αυτές οι συναντήσεις είναι σημαντικές εάν ε, μπορούμε να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και ε, για το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Συγκεκριμένα πράγματα. Δουλεύει ή δεν δουλεύει. Είμαστε ε, διασυνοριακά για να ε, απευθυνθώ στο θέμα της Φιλανδίας ε, Σουηδίας και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και έχουμε ε, σχέδια με αυτό το χώρο στάθμεσης, αυτό το σημείο ε, όπου θα βρίσκονται όλα τα προγράμματα και όλα όσα υπάρχουν μέχρι στιγμή είναι αυτό που θέλουμε να δουλέψουμε. βέβαια το τελικό αποτέλεσμα που στοχεύουμε είναι να έχουμε υπηρεσίες για τους πολίτες. Αυτές οι υπηρεσίες με που να είναι εντυπωσιακέ. Ε, στη Νέα Ζηλανδία λένε ότι θέλουν μια διαφανή κυβέρνηση, μια που να μην είναι ορατή αλλά να, υπάρχει, να υπάρχουν υπηρεσίε και να εξυπηρετούν του πολίτε όταν τι χρειάζονται. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε πλήρη ε, συμμετοχή των πολιτών. Αυτό θα το κάνουν τα κράτη-μέλη. Εμείς δεν έχουμε αρδομόδιότητες μέσα στα κράτη-μέλη, αλλά πολλά από τα επιτυχημένα κράτη-μέλη το κάνουν. Έχουν το περιβάλλον του εργαστηρίου, όπου βρίσκονται διάφοροι τομεί ε, και λύουν διάφορε διαδικασίε που πρέπει να απλουστευτούν. Ε, θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε, να απλουστεύσουμε, να αναθεωρήσουμε τι διαδικασίε έτσι ώστε να αφαιρέσουμε όλη την περιπλοκότητα και ε, ό,τι δεν χρειάζεται και ό,τι είναι περιττό. Να, δημιουργηθεί αυτό το αίσθημα του εργαστηρίου, όπου έχουμε ανατροφοδότηση από τους πολίτες και από την τρίτη ηλικία. Πώς συμμετέχει. Ναι, αυτό θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να εξαρτητοποιηθούν σε αυτό το στάδιο της ζωής, αλλά θα πρέπει να τους δοθεί και στήριξη ταυτόχρονα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το μοιραζόμαστε με κράτη-μέλη και έχουμε πολύ καλά παραδείγματα που έχουν, ε, ε, μας έχουν δείξει σε πολλές ε, περιπτώσεις, σε συνέδρια που έχουμε κάνει. Το ISA Square και τη ψηφιοποιημένη Ευρώπη πώς βλέπουμε το γεφύρωμα. Η κυριότερη ιδέα είναι να μπούμε στο πρόγραμμα DEP και να δούμε τις συνέργειες που υπάρχουν με άλλα προγράμματα. Να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέσα της Κομισιόν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ξέρει τι είναι τι. Μπήκαμε με ανοιχτό μυαλό για να βρούμε τις συνέργειες. Έχουμε μια σαφή περιγραφή του πώς θα συνεχιστεί το ΕΙΣΑ στο τετράγωνο, στο νέο πρόγραμμα. Ε, βέβαια δεν έχουμε ακόμη τα, την έκβαση και τα αποτελέσματα του προγράμματος του, της ψηφοποιημένης Ευρώπης και αυτό το κτίζουμε στους διαφορετικούς στόχους. Ε, τεχνητή νοημοσύνη, υψηλής απόδοσης, ε, υπολογιστές. Ε, όλα αυτά πρέπει να δουλεύουν μαζί για να υπάρχει ένα σετ από μέτρα που να λειτουργεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να στοχεύουμε κάτι που να ισχύει όλα τα κράτη-μέλη και στα προηγμένα, πολύ προηγμένα και υπάρχουν και στο βορρά και στο νότο και στην ανατολική στη δύση. Και για, θα πρέπει να δοκιμάσουμε ε, μαζί και να μοιραστούν οι εμπειρίες, αλλά μαζί επίσης με αυτά που δεν είναι τόσο προηγμένα. Θα πρέπει να στηρίξουμε τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, αυτές προβλέπουμε, για αυτούς που είναι πιο πίσω. Και ανάμεσα σε αυτά που έχουμε που είναι πολύ ε, ε, σημαντικά, είναι μέθοδοι αξιολόγησης. Δηλαδή, για να δει κανεί πού βρίσκεται με αυτές τις λύσεις, πόσο διαλειτουργικές είναι και από εκεί που είστε πώς μπορείτε να περάσετε στο επόμενο στάδιο και ε, έτσι ώστε να προχωρήσουν και τα λιγότερο προηγμένα μέλη. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης και ε, στο Single Digital Gateway. Εκεί έχουμε μια πρώτη εγγύηση για τους πολίτες για διαφορετικές διαδικασίες που υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη και ε, για παράδειγμα την Φόρμουλα Α1 <clears throat> ορισμένα πράγματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα όπου βρίσκεται κανείς, ε, δουλεύει, ζει, ε, σπουδάζει και αυτό προχωρεί πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό συμβάλλει το πρόγραμμα ΙΣΑ 2 γιατί γεφυρώνει τις εθνικές λύσεις με αυτό που χρειάζεται να γίνει ε, οικοδομώντας πάνω στην υποκείμενη αρχιτεκτονική, τη διασύνδεση ανάμεσα στο εθνικό και το ευρωενωσιακό επίπεδο λύσεων για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Βέβαια αυτό δεν είναι παρά μόνο το πρώτο βήμα. Είναι 20 διαδικασίες και πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Και επίσης δουλεύουμε με τους διάφορους τομείς, διότι πολλές από αυτές τις λύσεις είναι στις διάφορες ε, τομείς πολιτικής. Για παράδειγμα, ε, τα κοινωνικά ωφελήματα είναι στο χώρο της επασχόλησης. δουλεύουμε με τις γενικές διευθύνσεις να δούμε στα σχέδια εξυγχρονισμού τους πώς η Επιτροπή θα εξτάσει ε, τις επιχειρήσεις, πώς είναι τώρα, ποιες είναι οι προκλήσεις, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες ε, που ε, μας δίνει η ευφυής τεχνολογία για να περάσουμε ε, στο επόμενο στάδιο επίσης και στα θέματα πολιτικής. Και επίσης πανερχόμαστε και στα δεδομένα και στις τεκμηριωμένες αποφάσεις και την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Αυτά είχα να πω. Ε, χαίρομαι να ακούσω περαιτέρω εισηγήσει. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τι απαντήσει που δώσατε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας ευχαριστώ που μα εξηγήσατε τι συμβαίνει μέχρι τώρα, πώς μπορούμε την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη να τη βελτιώσουμε. Σας παρακαλώ βασιστείτε σε εμά και αν έχετε κάτι το συγκεκριμένο να ξέρετε πως θα συνεχίσουμε τις σχέσεις που έχουμε και το διάλογο που έχουμε και θα στείλουμε προτάσεις από τους συναδέλφους ενδεχομένου σε εσάς και στην ομάδα σας για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για να λειτουργούν καλά οι υπηρεσίε αλλά και υπέρ ε, του Ευρωπαίου Πολίτου. Σε 10 λεπτά θα έρθει η επίτροπο κυρία Γκάμπριλ. Θα έχουμε μία ώρα για να συζητήσουμε τα προγράμματα έρευνα και τα μελλοντικά σχέδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Parla Dear colleagues, uh, Συνάδελφοι, προτείνω να ξεκινήσουμε, να υποφεληθούμε πλήρως ε, της παρουσίας της Επιτρόπου Μαρία Καμπριέλ σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. Αν ε, είμαστε όλοι έτοιμοι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας και πάλι θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την κυρία Μαρία Γκαμπριέλ, Επίτροπο καινοτομία Έρευνα Πολιτισμού, Παιδεία και νέόλείας. Να πω ότι είναι η πρώτη επίσκεψη της Επιτρόπου Καμπριέλ στην Ήτρε μετά την ακρόασή της. Χαιρόμαστε που την βλέπουμε μαζί μας σήμερα. Ελπίζουμε να μάθουμε περισσότερα για την ε, τον συνεχισμένο σχεδιασμό του ορίζοντα Ευρώπης ε, και πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή και κάποια πράγματα και για τη νέα σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα τη έρευνα και ανάπτυξη. Θέλαμε να ε, συζητήσουμε επίση τι πρωτοβουλίε έρευνα και καινοτομία που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα εργασία τη Επιτροπή λόγω ε, ενός βάρη προγράμματος ε, και μας και της Επιτρόπου. Έχουμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας. Σας, λοιπόν, σας παροτρύνω να είμαστε όλοι αποτελεσματικοί, αποδοτικοί και να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αυστηρός μπορώ με τα χρονικά μας πλαίσια. Έχουμε όμως μία ώρα στη διάθεσή μας. Είναι αρκετός χρόνος να αγγίξουμε τα σημαντικότερα θέματα. Έχουμε επίσης ε, ένα κατάλογο ομιλητών για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη διεκπαιρέωση των εργασιών μας. Θα ξεκινήσω με κάποια εισαγωγικά ε, με την Επίτροπο. Θα κάνουμε επίσης ε, τις παρεμβάσεις των συντονιστών ή των αναπληρωτών τους και στη συνέχεια η Επίτροπος Γκαμπριέλ θα δώσει σύντομες απαντήσεις σε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και μετά θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος ε, με 12 συναδέλφους που είναι στο κατάλογο των ομιλητών και στο τέλος η κυρία Επίτροπος θα απαντήσει και σε εκείνες τις ερωτήσεις. Αν έχουμε βέβαια το χρόνο θα ε, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλους ε, ομιλητές που δεν είναι στον κατάλογο αλλά θα δυσκολευτούμε λίγο νομίζω. Άρα ξεκινάμε τώρα και δίνω αμέσως στο λόγο στην Επίτροπο Γκάμπριελ. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κριστιαν, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή, όπως είπε και ο Πρόεδρός σας, είναι ο πρώτος διαστρωμένος διάλογος που γίνεται στα πλαίσια της νέας ε, θητείας μου, ε, στη θέση της ε, Επιτρόπου για τα θέματα της αρμοδιότητάς μου και είναι πολύ σημαντικός για μένα ο διάλογος και τους επόμενους, τα επόμενα πέντε χρόνια θα ενισχύσω το διάλογο αυτό μαζί σας. Οι υπηρεσίες μου δίνουν ε, τις επαφές μαζί σας. Εγώ τους προέδρους και τους συντονιστές των δύο αρμοδίων επιτροπών ε, του συναντώ και εδώ και στο Στρασβούργο και χαίρομαι που συνεχίζονται αυτές οι ανταλλαγές. Και επιπλέον επειδή όλα αυτά είναι υπέρ των πολιτών, έτσι ώστε η πολιτική μας να είναι όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα επιτόπου. Θα ήθελα λοιπόν να σας μεταφέρω και κάθε επιτυχία στα νέα μέλη της Επιτροπής Ήτρε, όσους ε, πήραν τη θέση τους εφού αναχώρησαν οι Βρετανοί ε, συνάδελφοι και θα ήθελα ε, να μιλήσω μαζί σας για κάποιες πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο μου. Γι' αυτό θα μιλήσω για τρία θέματα Καταρχήν θα ξεκινήσω με τις προτεραιότητες, το Green Deal της ε, πίδελταπή μετά για τις νομοθετικές μου προτεραιότητες, Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνος, Διεθνή Συνεργασία, και πρόσφατη ε, ε, πρωτοβουλία για την βιομηχανική πολιτική, της μικρομεσαίας επιχειρήσεις και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως επίσης και το σχέδιο για την καταπολέμηση των καρκίνων. Και στο τέλος θα μιλήσω για το στρατηγικό σχέδιο και τις εταιρικές σχέσεις ως τρίτο κεφάλαιο. Λοιπόν, πολιτικές προτεραιότητες. Το έχετε δει και εσείς. Τις πρώτες 100 ημέρες η Επιτροπή Βαντερ Λάιν τήρησε τις υποσχέσεις της και κατέθεσε το Green Deal μία μόνη ανησυχία. Να διατηρήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος το χώρο της έρευνας ε, και της τεχνολογίας σε αυτή τη στρατηγική για να πετύχουμε τους στόχους μας. Γνωρίζουμε όλοι πως οι εθνικές πραγματικότητες είναι πολύ διαφορετικές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, το σημείο ε, άφηξης στο μυαλό μας ως ένα κοινό όρομα. Το σημείο αφετηρίας όμως είναι διαφορετικό για όλους. Και θέλω να συνεχίσω να ε, συνεργάζομαι με την Επίτροπο κυρία Φερέρα έτσι ώστε οι μηχανισμοί που προτείνονται και θα προτείνονται και μιλώ εδώ για το μηχανισμό της δίκαιης μετάβασης λαμβάνουν υπόψη τα απαραίτητα στο χώρο της έρευνα και τη καινοτομίας για να εξαλείψουμε τις διαφορές πι δέλτα πι 21-27 γνωρίζουμε πως ο χρόνος τρέχει. Σε 10 μήνες το πρόγραμμα Horizon ε, ε, Europe θα πρέπει να λειτουργεί. Και μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα πρικοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό, με τι φάκελο. Παραμένω αισιόδοξη αλλά επιφυλακτική. Θέλουμε ε, βορρά-νότο, ε, θέλουμε μικρομεσαίες, θέλουμε Νόμπελ και τεχνογνωσία και αυτά δεν θα τα πετύχουμε αν δεν έχουμε μια πολιτική έρευνας και καινοτομία στην Ευρώπη η οποία θα είναι γεμάτη περιεχόμενο. Ξέρω ποιες είναι οι δικές σας ε, φιλοδοξίες στον προϋπολογισμό, ξέρω τι θέλουν οι διάφορες κυβερνήσεις και σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Πρέπει να παραμείνουμε επιφυλακτικοί έτσι ώστε να υπερασπιστούμε τον κοινό μας στόχο ενός ρεαλιστικού και καλού προϋπολογισμού. Εδώ δεν μιλάμε για χρήματα απλώς, αλλά για επένδυση στο μέλλον και στο παρόν της Ευρώπης, κάτι που πιέζει. Είναι μια επίγουσα ανάγκη, θα το επαναλαμβάνω σε κάθε συνάντηση που έχω με τους ομολόγους υπουργούς, με τους πρωθυπουργούς, με τους υπουργούς οικονομικών και θα συνεχίσω και με, με τον Επίτροπο κύριο Χάν να συνεργάζομαι στενά. Στην επιστημονική κοινότητα μεταφέρω αυτό το μήνυμα καθημερινά και τους λέω συνεχίστε να προσπαθείτε στα πλαίσια των ε, κοινών μας ε, φωνών. Κάθε φωνή μετράει. Τους επόμενους μήνες, γιατί δεν νομίζω ότι την Πέμπτη θα τελειώσει το θέμα, ε, πρέπει να συνεχίσουμε να ακουγόμαστε. Τώρα, νομοθετικές πρωτοβουλίες, τρέχουσες και μελλοντικές. Καταρχήν, όπως είδατε και εσείς στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ιούνιο θα παρουσιάσω μια ανακοίνωση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και πώς θα τον αναζωπυρώσουμε, θα τον αναζωογονήσουμε. Είναι ένα θέμα πολύ προσφυλές, μια και για πρώτη φορά οι ευθύνε μου καλύπτουν και τις τρεις γωνίες του τριγώνου της γνώσης. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια νέα πνοή στο χώρο έρευνα στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε ε, τα επιστημονικά θέματα που προκύπτουν, ψηφιοποίηση, παγκοσμιοποίηση, μια βιώσιμη κοινωνία και βέβαια οι νέες προτεραιότητες όπως αυτή του Green Deal. Και γι' αυτό θα ήθελα να συνεργαστούμε πραγματικά έτσι ώστε ο χώρος αυτός να είναι πιο ανοιχτό σε όλους, πιο ελκυστικός πιο προσπελάσιμος σε καριέρα, σε αμοιβέ για τους ερευνητές μας, σε συνθήκες εργασίας και αυτά έτσι ώστε να ελαφρύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του brain drain και να μειώσουμε την κατάτμιση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά έρευνα στην Ευρώπη. Δεν θα το αφήσω αυτό από τα μάτια μου και στο Ζάγκρα πριν από μερικές μέρες είχα την ευκαιρία να ακούσω τον Φιλίπ Πουσκιά, πρώην Επίτροπο, να παρουσιάσει τον ε, απολογισμό των πρώτων 20 ετών της, ε, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να μιλήσω με τους υπουργού στο ε, Συμβούλιο σας και σας λέω πως υπό Γερμανική Προεδρία θα γίνει υπουργική διάσκεψη και εμείς θα αφιερώσουμε τις ημέρες μας ε, που μας συντηστοιχούν στην έρευνα και την καινοτομία το Σεπτέμβριο σε θέματα παρόμοια. Επίσης θα κάνουμε και ένα γύρο πρωτευουσών, έτσι ώστε να εξηγήσουμε ποιες είναι οι νέες μας φιλοδοξίες και κυρίως για να ακούσουμε ποιες είναι οι προσδοκίες των κρατών μελών, πώς μπορούμε μαζί να δημιουργήσουμε τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους μας. Για την διεθνή συνεργασία θέλω να πω δύο λόγια. Η Κροατική Προεδρία είναι πάρα πολύ φιλόδοξη για το Άστρο 12 και θα κάνει μία πρώτη στρατηγική συζήτηση στα πλαίσια ε, του Συμβούλου Ανταγωνιστικότητας 28 Φεβρουαρίου. Πολιτική βούληση είναι να συμφωνήσουμε εκεί και γι' αυτό η συζήτηση σήμερα είναι πραγματικά ε, καλή. Είναι 10 μέρες πριν το Συμβούλιο και για μένα είναι σημαντικό να έχω ακούσει τη δική σας άποψη μέχρι τότε. Προφανώς η συμφωνία για το άρθρο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια συμφωνία έτσι ώστε και εμείς από την πλευρά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις, τις διερευνητικές σε τεχνικό επίπεδο με τρίτες χώρες. Και τέλος, πάντα νομοθετική μας προτεραιότητα είναι τα κάτωθη τρία θέματα. Τεχνητή νοημοσύνη, καταρχήν, θα εγκριθεί αύριο. Και ως πρώην επίτριος για τα ψηφιακά φαντάζεστε πόσο σημαντική είναι η πρωτοβουλία αυτή για μένα. Πάντα ήμουν υπέρ του να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρος και σκαπανέας στο σημείο αυτό και η τεχνολογία να συνοδεύει τα ανθρώπινα όντα και πουδενή να υποκαταστήσει αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν στην υπηρεσία του ανθρώπου που θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην υγεία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, Βλέπετε λοιπόν είναι θέματα τα οποία είναι κομμάτι του νέου Horizon Europe δεν θέλω εγώ μια τεχνητή νοημοσύνη που θα ε, αποφασίζει αντί για εμάς. Στις συζητήσεις λοιπόν που κάνουμε ε, με τον Επίτροπο κύριο Μπρετό τα θέτω αυτά και είναι επίσης στρατηγικό το θέμα γιατί είμαι πεπισμένη πως μια προστασία περιβάλλοντος αποτελεσματική, μια στεναρή βιομηχανική πολιτική μπορούν να συνδυαστούν είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αποτελεσματικό τρόπο για να δουλεύουν καλά. Και είμαι πολύ ικανοποιημένη που ήδη φαίνονται τα πρώτα θετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα του Συμβουλίου ε, καινοτομία. αυτή η μονοθυριδική υπηρεσία, το one-stop shop, έτσι ώστε να μπορούν να απευθυνθούν εκεί οι νεοφυείς υπηρεσίες και οι μικρομεσαίες για να λάβουν χρηματοδότηση. Επιβεβαιώνω λοιπόν πως οι φιλοδοξίες μας είναι να αλλάξουμε μέσω του Συμβουλίου Καινοτομίας τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την καινοτομία και να αποτελέσει τη βάση για συμφωνίες στην Ευρώπη έτσι ώστε παγκόσμια να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από μένα. Δεν μας λείπουν οι startups στην Ευρώπη. Έχουμε περισσότερες από ό,τι στις είπα. Εμείς δεν ξέρουμε πώς να τις βοηθήσουμε να μεγαλώσουν και να ανεξαρτοτοποιηθούν. Εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος της προσπάθειάς μας. Και θα ήθελα να μιλήσω και για μια σειρά θεματικών προτεραιοτήτων, το strategic planning, στρατηγικό σχεδιασμός. Είδατε το Γενικό Διευθυντή κύριο Πακέ, και είναι μια χωρίς προηγούμενο προσπάθεια συνδημιουργία. Σήμερα το πρωί ήμουν στην Επιτροπή Περιφερειών για να συνεχίσω εκεί με τη διαδικασία τη συζήτηση από τον ιδιωτικό κλάδο, από την κοινή γνώμη και από τον επιστημονικό κόσμο για να προχωρήσουμε χέρι-χέρι και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Είμαστε τη στιγμή της ε, σύνταξης του σχεδίου για τη νομική βάση του Horizon Europe. Έχουμε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τα όσα ακούσαμε ως σχόλια και όλα αυτά προσπαθούμε να τα συγκεράσουμε. Θα γίνει και μία ακρόαση ε, δημόσια για τα θέματα που με αφορούν. Τώρα, να σας πω τώρα πως για το θέμα των ε, εκπομπών θα πρέπει να δούμε τι λέτε εσείς και τι λένε οι πολίτες μας. Γιατί θα πρέπει οι στόχοι αυτοί να γίνουν κομμάτι και τμήμα των ίδιων των πολιτών για να πετύχουν, για τις εταιρικέ σχέσεις. Θα πρέπει εδώ να εξορθολογήσουμε. Έχουμε 120 και θα πάμε σε 44. Θα δούμε με τα κράτη-μέλη πώς μπορούμε να δώσουμε κάποιο περιθώριο. Για μένα όμως είναι σημαντικό γιατί μαζί μας θα πρέπει να συντάξουμε για τις εταιρικές αυτές σχέσεις ε, να δημιουργήσουμε τα κριτήρια. Να είναι συνεκτικές, να, να έχουμε συνέργεια στις προσπάθειες αυτές, ε, να ακολουθούμε την, κοινωνική, την κοινή λογική. Η δική σας ε, πρόταση για τον OIT θα βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε ένα νέο κικ, αλλά ακόμα πιο ε, διάφανο, ακόμα καλύτερο από ό,τι στο παρελθόν. Να σας πω πως ξεκινήσαμε και με μία επιπτωσιολογική μελέτη ε, για τους 13 υποψηφίου για τις εταιρικέ σχέσεις στα πλαίσια του 185 και 187. Η μελέτη αυτή βιωσιμότητας θα μας επιτρέψει στο δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς να προχωρήσουμε με προτάσεις νομοθετικές για το θέμα αυτό. Κλείνω εδώ για να συζητήσουμε με μεγάλη άνεση χρόνου Θέλω εδώ να σε ευχαριστήσω και πάλι γιατί είναι μήνες τώρα που δουλεύουμε μαζί και συμμεριζόμαστε το ίδιο όραμα να επιβεβαιώσουμε δηλαδή πως η παιδεία, η εκπαίδευση, η καινοτομία, η έρευνα είναι οι προϋποθέσεις, η εκ των όνου άνευ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομία. Είναι ο μοναδικός τρόπος να πετύχουμε την μετάβαση, την οικολογική, κοινωνική και οικονομική που επιδιώκουμε και θα χρειαστώ να συνεχίσετε να είστε έτσι ενθουσιώδης, έτσι γεμάτοι ιδέες, έτσι υποστηρικτικοί προς τα εμένα και θα συνεχίσω να έρχομαι εδώ στο δυνατόν πιο συχνά. Δίνω τώρα το λόγο στους συντονιστές από τις πολιτικές ομάδες. ΕΛΚ, η κυρία Καρβάλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Επιτροπέ, για την παρέμβασή σας και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια μικρή μου τοποθέτηση και μετά ε, θα κάνω δύο ερωτήσεις. Η τοποθέτησή μου αφορά τον προϋπολογισμό και ε, στο γεγονός ε, ότι μπορείτε να βασιζόσαστε σε εμά για να επενασπιστείτε τον προϋπολογισμό που έχετε καταθέσει για το πρόγραμμα Horizon. Βλέπουμε λοιπόν όλο και περισσότερο πολλές ανακοινώσεις ε, που προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις ε, που να βασίζονται ε, στο πρόγραμμα Horizon δημόσιες πρωτοβουλίες, τεχνητή νοημοσύνη. Άρα δηλαδή το πρόγραμμα Horizon θα είναι πολύ σημαντικό για την Πράσινη Συμφωνία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ψηφιοποίηση. Άρα στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να προβλέψουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να προκύψουν και τα αναμενόμενα από τον τομέα της ε, έρευνας και της ε, τεχνολογίας. Γιατί ε, από εκεί θα προκύψουν οι λύσεις για την πράσινη οικονομία και για τη μετάβαση, πράγματα που χρειάζεται η οικονομία μας. Και θέλω να ρωτήσω, μήπως μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι στο θέμα των αποστολών που υπάρχουν. Ε, προβλέπονται καινούριε. Και πότε υπάρχουν προγράμματα για νέες αποστολές. Επίσης, όσον αφορά τις ε, συνεργασίες, μας είπατε ότι υπάρχει κάποια αξιολόγηση για τις ε, συνεργασίες ε, φαντάζομαι αναφέρεστε στις ε, θεσμοθετημένες ε, συνεργασίες. Κατά τα άλλα, πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο. Μιλήσατε για την νομοθετική εργασία. Μέχρι τώρα, ο ερευνητικός χώρος στην Ευρώπη ήταν περισσότερο μία έννοια, δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει νομοθεσία, γιατί υπάρχουν τα κράτη-μέλη ε, τα οποία καλούνται να δραστηριοποιηθούν στο θέμα της ψηφιοποίησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας έχουμε στην Επιτροπή μας. Ταυτόχρονα θα ήθελα να να σε εκφράσω την ανησυχία που έχουμε, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι στις 20 Φεβρουαρίου θα έχετε μια σημαντική ε, παρουσία στο Συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός, το ΠΔΠ, το εμείς ε, σήμερα συζητάμε τον προϋπολογισμό για τον ορίζοντα Ευρώπη. Εμείς στηρίζουμε την θέση του Πρόεδρου Σασόλη που ε, θεωρεί ότι δεν είναι υπαρκής επαρκή τα κονδύλια για, στο ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ και θα εξηγηθώ μόνο για το θέμα του ορίζοντα. Για τα 80,9 δις ε, αυτό θα σημαίνει κύριε Επίτρεπε τα ακόλουθα θέματα. 10 ε, δις πτώση σημαίνει ε, πτώση κατά 110 δις δολάρια σε 25 χρόνια. Ε, μείωση θέσεων απασχόλησης μέσα στο 2040. 300 ερευνητικά προγράμματα που θα χαθούν 1.700 σχέδια λιγότερα στο, θέμα, ε, στο πρόγραμμα Marie Curie, λιγότερα ερευνητικά προγράμματα και συνεργασιακά προγράμματα, 1.000 ε, επιδοτήσεις λιγότερες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 50.000 ερευνητές που θα λάβουν λιγότερα κονδύλια, 11.600 ε, λιγότεροι ερευνητές που θα έχουν πρόσβαση σε υποδομή έρευνας. 28.000 ε, peer review publications θα χαθούν, ε, απώλεια 900 ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, θα χάσουμε επίσης 7.000 πρωτότυπα και 12.000 δραστηριότητες δοκιμασιών και 500 κλινικές δοκιμές που θα πάνε χαμένες επίσης στον ερευνητικό τομέα. Είναι λυπηρό, είναι αδύνατο και δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνεται αυτές οι προτεραιότητες που γνωρίζουμε όλοι ε, και πώς θα βρεθούν αυτά τα κονδύλια. Και ε, θα ήθελα να πω ότι στις ανταλλαγές που γίνονται, για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί η Κομισιόν με το Κοινοβουλίο και δεν είμαστε ε, αντίπαλοι. Αντιθέτω, ο κοινό σκοπό είναι να ε, πετύχουμε το καλό για αυτού που περιμένουν από την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα για του ερευνητέ και για την ερευνητική δραστηριότητα για το πιλωτικό πρόγραμμα. Περιμένουμε για τα blind evaluations να δούμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και να δούμε τα αποτελέσματα του πιλωτικού προγράμματος και στην διεθνή συνεργασία είχαμε μια πρώτη συνάντηση με τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης για την ε, ε, ε, διεθνή συνεργασία. Ζήσαμε να έχουμε ad hoc συναντήσεις για ένα πρόβλημα πολύ ευαίσθητο, το οποίο θέλουμε να χειριστούμε με κάθε προσοχή. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μην δεχτείτε ε, αυτές οι ε, διαπραγματεύσεις να είναι ιδιωτελείς, διότι εκεί θα έχουμε ένα πρόβλημα όταν φτάσουμε σε άλλες χώρες και άλλες καταστάσεις και θα έχουμε ένα ε, ολοκληρωτικό πακέτο, να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα ποσά και τα κονδύλια και ποιο είναι το σωστό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχετε επιτυχία και να έρθετε με τα απαραίτητα κονδύλια για την έρευνα. Ευχαριστώ κυρία Νίκα και κυρία Τζαμπαϊόβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Νομίζω όλοι θα έχουμε μια κοινή γραμμή σε ορισμένα θέματα όπως είναι ο προϋπολογισμός. Βέβαια περιμένουμε με ενδιαφέρον ε, τις αντιδράσεις των κρατών μελών ε, από ε, τις προτάσεις του Σαρ Μισελ, αλλά όπως γνωρίζετε η γραμμή του Ευρωκοινοβουλίου είναι σαφέστατη. Η έρευνα και η καινοτομία έχει προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη, γι' αυτό ζητάμε για περισσότερα κονδύλια και σα ζητάμε να κρατήσετε ισχυρή θέση εκεί. Αυτό είναι ένα πράγμα είναι σημαντικό ε, λόγω της σημασίας του ορίζοντας στις νέες προτεραιότητες πολιτικές της Κομισιόν, πώς θα το σχηριστεί η Κομισιόν, πώς θα αναθεωρήσει την θέση της για την εσωτερική ε, ανάλυση του προϋπολογισμού για αυτό το κεφάλαιο. Διότι ε, πριν από δύο χρόνια οι προτεραιότητες ήταν διαφορετικές με την προηγούμενη Επιτροπή. Σήμερα συζητάμε καθημερινά για θέματα τεχνής νοημοσύνης, πράσινης συμφωνίας. Ήταν διαφορετικό πριν από δύο χρόνια με τις προτάσεις της προηγούμενης Επιτροπής. Πώς το βλέπετε εσείς και πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό, ίσως μαζί σε αυτές τις νέες προτεραιότητες της νέας Κομισιόν. Και δεύτερο σημείο. Είναι πιο η, οριζόντια η προσέγγιση. Θα πρέπει να δούμε συνέργειες, διεθνή συνεργασία. Ε, βιομηχανική πολιτική αυτή καθ' αυτή. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία και θα χρειαστούμε το συντομότερο δυνατόν να έχουμε οριζόντια προσέγγιση σε κοινέ διατάξεις ε, ανάμεσα στις προτεραιότητες της Ήτρα και της Ρέτζη, για παράδειγμα. Θα πρέπει να δουλέψουμε μαζί σας, θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στις επιτροπές. Και τέλος, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είπατε κάτι, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι και τόσο συγκεκριμένα όσο θα έπρεπε να ήταν η αντίδρασή μας προς τους πολίτες. Βέβαια θα διεξαχθεί σύντομα αυτή η συζήτηση για τη στρατηγική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά φοβάμαι ότι ήδη έχουμε βιώσει ε, στα τελευταία προγράμματα ότι δεν υπάρχει αρμόδια στελέχωση στις ε, μικρομεσαίες για μεγάλα έργα όπως είναι ο ορίζοντας και είναι ε, περίπλοκες οι ε, διαδικασίες είναι ε, διαφορετικό σε κάθε παρπιστήμιο, σε ερευνητικό κέντρο. Πώς διασφαλίσουμε λοιπόν την πρόσβαση των μικρομεσαίων σε μεγάλες προσκλήσεις ενδιαφέροντος και μεγάλα προγράμματα καινοτομία, Γιατί ε, στις ημέρες έρευνα και καινοτομίες μόνο οι μεγάλοι παίκτες τελικά ε, παρευρίσκονται εκεί. Θέλουμε και την παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θέλουμε κάτι πιο συγκεκριμένο ειδικά εξειδικευμένο γι' αυτό. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ε, του ΑΕΔ, κυρία Έλενα Ρίτσι. Ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Ε, το πρόγραμμα Horizon Europe. Εγώ είμαι σκιώδης ε, για την πολιτική ομάδα ID και θα ήθελα να έχω κάποιες ε, διευκρινήσει. Ε, γιατί οι ερευνητές είναι νέοι και σε επισφαλή θέση απασχόλησης. Θέλω λοιπόν να πω το εξή. Η έρευνα και η τεχνολογία χρειαζόνται ιδέες, ε, χρειάζονται καινοτομία. Όμως εδώ ε, περίζουν τα κονδύλια και το χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου ε, το χρονικό διάστημα ίσως να μην φτάνει για να επιτύχει κανείς τόσο υψηπετής στόχους. Ίσως θα, πρέπει να κινητοποιηθούν επενδύσεις μέχρι και ένα 3 ευρώ, ίσως και περισσότερο. Ανταπτού η Κομισιόν θα διαθέσει 6,5 δις από ό,τι ακούσαμε. Τα υπόλοιπα που θα τα βρείτε ε, Πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα ε, εξασφαλίζουν στους πολίτες ότι τα προγράμματα προχωράνε. Δεν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές καλές προθέσεις αλλά πολύ λίγες πράξεις. Ένα μεγάλο κομμάτι ε, των προγραμμάτων και των κονδυλίων θα διοχετευτεί για την κλιματική αλλαγή. Τα υπόλοιπα κονδύλια πώς θα καταναμηθούν, μήπως έχετε κάποια ιδέα για την κατανομή των υπολείπων κονδυλίων. Και μία ερώτηση για τις εταιρικές σχέσεις. Πιστεύετε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια νέα σχέση ανάμεσα στις εκπομπές και τις συνεργασίες και εάν ναι, πώς θα πρέπει όλα αυτά να διοχετεύονται στο προπολογισμό. ποιε είναι οι νομοθετικέ διαδικασίε για κάθε μορφή συνεργασία, μήπω έχετε υπολογίσει και τι επιπτώσει από το Brexit στι συνεργασίε και αν ναι, πώς. Κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι όσον αφορά το θέμα των αποστολών. Εκεί υπάρχει έτσι μια γενική ε, αχλή, θα έλεγα. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, να μην ξεχνάτε ότι απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες οφείλουμε όχι μόνο απαντήσεις, αλλά και αποτελέσματα. Εμείς ως ομάδα ανησυχούμε πάρα πολύ, γιατί βεβαίω και συμμεριζόμαστε το ότι είναι σημαντική η έρευνα και η καινοτομία για το μέλλον, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται ε, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Η Επιτροπή ε, ε, είδαμε ότι πολλές φορές ε, μπορεί να στείλει την οικονομία σε αδιέξοδο και προφανώς και τις κοινωνικές σχέσεις. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθησυχαστικά σημάδια. Παρόλα αυτά ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα μπορέσει να μας πείσει με την ιδιότητά της του συνομοθέτη. Προς το παρόν δεν έχουμε δεχτεί τέτοιου είδους μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, ε, ο κύριος Νταλούντε, εκ μέρους των ε, Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά και της προηγούμενης θητείας είχα την τιμή να είμαι σκιώτη ηγητής ε, της ομάδας ε, Renew και πρέπει να σας πω ότι αυτό που μας απασχολούσε πάρα πολύ ήταν το mainstreaming. Το 35% βέβαια ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρό. Ε, πάρα πολλοί ζήτησαν 50% όχι μόνο οι πράσινοι και άλλοι, αλλά επίσης και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ, πανεπιστήμια και ευρωπαϊκές εταιρείες που ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτή την πράσινη μετάβαση. Το 50% της συμπερίληψης διάσταση του κλίματος στα προγράμματα, αυτό το συζητήσαμε στο Παρίσι και είπαμε ότι έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Πρώτη ερώτηση. Το Horizon Europe προτάθηκε ε, ως ένα πρόγραμμα το οποίο ε, έχει τύχει παλαιότερη διαπραγμάτευση και ρωτώ οι νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς θα επηρεάσουν ε, τον, τον νέο σχεδιασμό και πώς όλα αυτά θα φανούν στα προγράμματα του 2021 και 2022. Δεύτερη ερώτηση. Στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Ιανουαρίου και με την ομάδα για το Horizon, ο ε, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει πάνω σε μια στρατηγική ε, που να μπορεί να εφαρμοστεί. Ε, πότε λοιπόν θα μας δώσετε αυτή τη στρατηγική. Και τελευταία ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να διασφαλίσει ότι ό,τι απομένει από τον προπολογισμό του Horizon ε, δεν θα δαπανηθεί για δραστηριότητες ε, οι οποίες βλάπτουν τις ε, φιλοδοξίες μας ε, για το κλίμα. Ο κύριος Τωσανόφσκι εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, αγαπητή κυρία Επίτροπε, να ξεκινήσω κι εγώ με τις ευχαριστίες μου που για μια φορά ακόμα είστε εδώ και συζητάτε τα θέματα αυτά μαζί μας. Στην εισαγωγή που κάνατε, μας είπατε πως μετά από την έναρξη της νέας θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρώτο θέμα ήταν το Green Deal. Ένα από τα εργαλεία τα οποία προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συζήτηση έχει γίνει είναι το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση που θα πρέπει να βοηθήσει να ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες στις αλλαγές που θα γίνουν και τις οποίες θα χρειαστεί να περάσουν κάποια ε, κράτη ε, στις αλλαγές που θα κάνουν στην οικονομία τους, στην ε, μείωση της χρήσης του άνθρακα κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς θα πρέπει να συνδέσουμε αυτό το Ταμείο της Δίκαιης Μετάφασης και το Horizon Europe το έχουμε συζητήσει πολύ εδώ με τους συναδέλφους και ακόμα και με τους σκιώδεις και εμείς θέλουμε εδώ κάποιες δραστηριότητες να τις εντάξουμε και πιο συγκεκριμένα, εσείς πολύ σωστά είπατε πως υπάρχουν ιστορικές, γεωγραφικές, ε, πολιτιστικές ε, διαφορές μεταξύ περιοχών της Ευρώπης και χωρίς καινοτομία, γνώση, τεχνολογία αυτές οι αλλαγές θα μείνουν στα λόγια και δεν θα καταφέρουμε να τις μεταφρέσουμε σε πράξεις. Είπατε λοιπόν θα πάψουμε να εκμεταλλευόμαστε τον άνθρακα. Ωραία. Αν όμω η τεχνολογία, η επαναστατική αυτή, την οποία εμείς ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι να τα κάνουμε, θα μείνουμε σε ευχολόγια για το μέλλον, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει εξυπέραστα προβλήματα. Εσείς λοιπόν τι πιστεύετε, ποιε είναι οι συνέργειες μεταξύ της έρευνες και του Horizon ε, και του ε, Ταμείου για την ε, δίκαιη μετάβαση, γιατί είναι σημαντικό να το δούμε, μια και υπάρχει πάντα και ένα ενδεχόμενο ρίσκο. Ο κύριος Μποτέγκα, παρακαλώ, είναι ο τελευταίος στον κατάλογο. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Επίτροπε, για τα σχόλια που κάνατε. Εγώ για να μιλήσω γρήγορα δεν θα επανέλθω στο θέμα του προπολογισμού. Όλοι συμφωνούμε πως φιλοδοξία χωρίς προϋπολογισμό δεν σε πάει μακριά. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι πιστεύετε και για την ε, συνέπεια των όσων κάναμε. Εσείς μιλήσατε για ένδια, για δυσκολία, για βεβαιότητα. Να σας πω πως για πρώτη φορά η Ιταλία στην, ιστορία της κατάφερε να προσλάβει ε, με πραγματική σύμβαση, μία ερευνήτρια, ε, μία ερευνήτρια η οποία 13 χρόνια ζούσε με ε, περιορισμένου χρόνου συμβάσεις, με μεγάλες δυσκολίες. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν, στην ε, μάχη κατά της αστάθειας επαγγελματικής των ερευνητών, τι όπλα θα χρησιμοποιήσετε για τη βιομηχανία τώρα στα ερευνητικά προγράμματα. Θέλω να μου πείτε τι θα συμβεί και πώς θα μεταφούμε σε μια καθαρή τεχνολογία. Στη σιδηρουργία, για παράδειγμα. Θα χρησιμοποιήσουμε πράσινο υδρογόνο. Επίσης, σε αυτό το επίπεδο ποιες είναι οι προτεραιότητες. Θα είναι στο 35% της ε, χρηματοδότησης για το κλίμα. Είναι κάτι πιο διευρυμένο ή θα είναι στις προτεραιότητες τις οποίες θα καταθέσετε. Και πώς είστε βέβαιοι πως τα πλέον εκτίματα θα τα χαρεί ολόκληρη η κοινωνία και δεν θα τα καπαρώσουν κάποιοι ιδιώτες ε, σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μποτέγκα. Έκλεισε λοιπόν ο πρώτος γύρος ερωτήσεων στα πλαίσια του διαλόγου μας. Θα ζητήσω τώρα από την Επίτροπο να δώσει κάποιες απαντήσεις. Αλλά σας παρακαλώ πολύ πέντε λεπτά. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Αλλά έχουμε ακόμα 12 συναδέλφους και θέλουμε να τους ακούσουμε όλους. Έχουμε λοιπόν ερωτήσεις για τον προϋπολογισμό, αλλά έχουμε και ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους. Για μια φορά ακόμα μιλήσατε στην ανάγκη να υπερασπιστούμε τον προπολογισμό μας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το ακολουθήσουμε και όπως είπατε και εσείς, εγώ από πλευρά μου δεν θα, βάλω, δεν θα τα παρατήσω, δεν θα τα βάλω κάτω. Θα κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε οι φιλοδοξίες μας να έχουν τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να τις πετύχουμε για τις διάφορες ερωτήσεις. Κυρία Καρβάλιο, σας ευχαριστώ για τις εταιρικέ σχέσεις. Ναι, η επιπτωσιολογική μελέτη Impact Assessment τρέχει. Είμαστε καλά σε σχέση με τους χρόνους μας. Για τη συγχρηματοδότηση, για μας το πιο σημαντικό είναι η μείωση αυτών των εταιρικών σχημάτων να μειωθούν. Σχημάτων. Θα φτάσουμε τα 44 από τα 120 και προσπαθούμε τα νέα κριτήρια που έχουμε θέσει να είναι συνεπή να μην έχουμε επικαλύψεις, να εστιάζουν στα αποτελέσματα και στα παραδοτέα και να κλείσει η δουλειά που αυτή τη στιγμή τρέχει. Η γνώμη του Κοινοβουλίου είναι βεβαίως καλοδεχούμενη. Θέλουμε για μια φορά ακόμα να είμαστε αποτελεσματικοί και να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να προχωρήσουν στο σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας της Ένωσης. Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ αμέσως νομοθετικό έργο, αλλά μας έδωσε το άνοιγμα αυτό ήδη η συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, οπότε ας αρπάξουμε την ευκαιρία. Και ξέρω πως στις δικές παρεμβάσεις είπατε πως οι αμοιβέ, οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων στην έρευνα είναι σημαντικές. Εμείς θα πούμε πόσο σημαντικό είναι τα ταλέντα μας να μένουν στην Ευρώπη, χρειάζεται. Εμείς θα πούμε ότι χρειάζεται να τους δώσουμε κίνητρα. Πρέπει στα όταν κλείσει η τρέχουσα διαδικασία να ξεκινήσουμε κάποιες συζητήσει για το τι σημαίνει Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και τότε να συνταχθεί το Κοινοβούλιο μαζί μας και στο γύρο του προεδρευουσών που θα κάνουμε και ε, να δούμε στην ανακοίνωση του Ιουνίου ποιε θα είναι οι βάσει για συστάσεις συγκεκριμένε που θα μα επιτρέψουν να ξεπεράσουμε την απλή αγορά ε, στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση αυτή τη στιγμή όπως θα θέλαμε εμείς να φαίνεται. Και νομίζω ότι θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Αν οι συστάσεις αυτές στηριχθούν, γίνονται εκτεσθετικά, θετικά, τότε ναι, εγώ να πάω και πιο μακριά και το λέω και πάλι. Εγώ δεν βρήκα οι υπουργοί να έχουν αντιρρήσει. Στην πρώτη συζήτηση πριν από 15 μέρες στο Ζάγκρεπ ήταν πολύ ενθαρρυντικά τα πράγματα για την ανάγκη που υπάρχει να ενημερώσουμε, να ε, αναζωογονήσουμε αυτό το χώρο στην Ευρώπη. Τώρα, για την αξιολόγηση των project, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκα για τα νούμερα που δώσατε. Θα πρέπει να τα διαδώσουμε απλώς. Θα πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι στην Ευρώπη. Γιατί διαφορετικά έχουμε την τάση να ξεχνάμε και μετά να πούν πως η εξολόγηση των project θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, η ομάδα μου και εγώ έχω δώσει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, είναι σημαντικό. Τώρα, για το πώς θα κάνουμε ανακατανομή μέσα στα κεφάλαια. Δεν έχουμε μιλήσει για τέτοιου είδους κλιμάκωση. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, το Green Deal, αλλά στον προϋπολογισμό του Horizon Europe έχουμε και εργαλεία που είναι τα απαραίτητα ε, και μπορούμε να εντάξουμε. Το 35% του προϋπολογισμού στο Horizon Europe θα αφιερωθεί στην ε, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και οι υποθέσεις αυτές θα ειδωθούν και στα πλαίσια του Green Deal. Αυτά θα τα κάνω και θα τα δούμε πριν κάνουμε νέες προτάσεις και για την τεχνητή νοημοσύνη. Μην ξεχνάτε, έχουμε το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη Δυόμιση δις. Δυόμιση δις. Θα φέρουν τη διαφορά. Και μετά βλέπουμε. Είμαι πολύ ξεκάθαρη. Τα χρήματα του Horizon Europe θα χρησιμοποιηθούν μόνο όπου είναι απαραίτητο και μόνο εκεί που υπάρχει προστιθέμενη αξία. Έχουμε το πλαίσιο με την κατάλληλη ευελιξία για να προσαρμοστούμε στις νέες προτεραιότητες. Επίσης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό και επιμένω για το ρόλο που έχει το Συμβούλιο καινοτομίας, Το 70% του προπολογισμού θα πάει στις μικρομεσαίες. Θέλουμε να επενδύσουμε με τα δύο σχήματα και κυρίως με τον επιταχυντή. Και εκεί να σας πω πως ένα από τα θέματα τα οποία έθεσε ο κύριος Ντελούντε, Θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε project τα οποία δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και γι' αυτό αποφασίσαμε στην επόμενη πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομία που θα προκηρυχθεί ε, το Μάιο, 300 εκατομμύρια μόνο για νεοφυείς και μικρομεσαίες που θα επενδύσουν σε πράσινη τεχνολογία. Θα το παρακολουθήσουμε στενά και θα πρέπει εδώ να προσθέσουμε τα skills, τις δεξιότητες. Το είπατε, συνάδελφε Λαμπάζοβα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κενά, προκλήσεις θα πρέπει να έχουν περισσότερα εργαλεία και εκεί πια δυσκολεύει πολύ η κατάσταση και πήγε να συνεργαστούμε όχι μόνο με τον κύριο Μπρετόν αλλά με τον επίτροπο κύριο Σμιτ έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και εγώ είμαι έτοιμη να οργανώσω και μεικτή συνάντηση με τον Επίτροπο κύριο Μπρετόν έτσι ώστε να φωτίσουμε τα ζητήματα τα οποία εσείς θέσατε, να μην έχουμε επικαλύψεις και να μην σπαταλάμε πόρους. Και κάτι το οποίο για μένα είναι ιδιαίτερα προσφυλές είναι οι συνέργειες μεταξύ των υπολείπων και δεν σας κρύβω πως το Δεκέμβριο ξεκίνησε μια συνάντηση ε, με με τους επιτρόπους την κυρία Φερέρα και τον κύριο Σμιτ ε, κάθε τόσο για να βρούμε ε, Του κατάλληλο τρόπο για να μην μείνουν όλα αυτά ε, λόγια στο χαρτί. Μετάβαση ταμείων, μεταφορές, ε, κοινωνικό ταμείο, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορούμε να μετακινούμε χρήματα και για τους νέους ερευνητές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, τι θα κάνω την επόμενη εβδομάδα. Για την υποτροφία Marie Curie θα προτείνω η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει το σύνολο του ποσό για τους διδάκτορες και για τους όσους κάνουν ε, μεταδιδακτορικό ε, και να μειώσουμε και την ηλικία για να αυξηθεί κατά 20% η συμμετοχή. Δεν μιλάμε για θαύματα, μιλάμε για μικρά συγκεκριμένα βήματα τα οποία παρουσιάζω έτσι ώστε να δώσουμε το μήνυμα πως οι ερευνητέ στην Ευρώπη στηρίζονται και έχουν μέλλον. Περνούμε <clears throat> πάρα αυτά στο δεύτερο γύρο. Κυρία Σπυράκη, για ένα λεπτό, παρακαλώ να κρατούμε το χρόνο μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε εδώ. Όπως είπατε κι εσείς, ο ορίζοντας είναι μια επένδυση για το μέλλον, αλλά στη θητεία σας Εκτός από επένδυση για το μέλλον, θα πρέπει να περιλάβουμε και την νεολαία. Θα ήθελα να δω κατά πόσο ο κανονισμός θα περιορίσει τον ελεύθερο, τον ελεύθερο λόγο. Και η ερώτηση είναι, η Επιτροπή είναι έτοιμη να ενθαρρύνει καινοτόμο εφαρμογή, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τις οικογένειες και για μας ως γυναίκες, ως μητέρες. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ ε, κύριε Επίτροπε. Κοιτάξτε, ε, όταν ε, μιλάμε για την Πράσινη Συμφωνία, μιλάμε για την έρευνα, γιατί όπως είπατε και εσείς, είμαι πεπισμένη ότι η κλιματική ουδετερότητα αυτό σημαίνει ένα τεχνολογικό άλμα, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει ίσως να υπάρχει και μια διαφορετική ε, βιομηχανική ε, στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει με την Πράσινη Συμφωνία να ξέρουμε τι επιθυμούμε και πώς μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας και με την έρευνα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για να θέσουμε λιγάκι και το θέμα του Horizon στο παιχνίδι, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Πώς μπορούμε, πώς μπορείτε να έχετε εσείς ε, το δικό σας το χαρτοφυλάκιο τέτοιου είδου θέματα, γιατί πρέπει να ρίσουμε το θέμα των αποστολών και των συνεργασιών. Και ακόμα και αν μερικές φορές ε, ε, υπάρχουν όρια, και παρόλα αυτά όμως πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αποφασισμένοι ε, για να μην υπάρχει αυτή η αποκοπή, οι μένα ασχολούνται με τα α και να μην υπάρχει συνεργασία. Η κυρία Μιχαήλοβα. Κύριε Επίτροπε, θα μιλήσω βουλγαρικά. Ε, πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Ε, εσείς ε, αναφερθήκατε στην σωστή χρήση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη η επιστημονική έρευνα δεν προχωράει γρήγορα και σε άλλες πάλι, πάλι περιπτώσεις η έρευνα ε, προχωράει πολύ περισσότερα, πολύ πιο γρήγορα. Το ίδιο ισχύει και για την καινοτομία. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε κάποιες ε, γέφυρες. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συμπεριληφθούν χώρες με περιορισμένη συμμετοχή. Από ό,τι φαίνεται, στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, πρέπει να είμαστε περισσότερο ευέλικτοι. Πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις χώρες που το χρειάζονται. Αγαπητοί κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε για όλα αυτά που είπατε σήμερα, πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι ε, κάνετε μία από τις σημαντικότερες ερωτήσεις, δηλαδή πώς μπορούν να ε, αναπτυχθούν περαιτέρω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πολύ συχνά ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν ότι υπάρχουν εμπόδια όταν ετούνται κονδύλια από το πρόγραμμα Horizon. Επίσης, πολλές φορές λένε ότι δεν αξίζει τον κόπο να ζητήσουν κονδύλια, πάρα πολλές ε, μένουν ε, πιο πίσω, παραμελούνται. Ε, γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το να ετηθεί κανείς κονδύλια από το πρόγραμμα Horizon θα είναι πολύ πιο εύκολο. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και εγώ ε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ανησυχώ πάρα πολύ για τον προπολογισμό του Horizon. Δεν θα ρωτήσω για εκεί, θα ρωτήσω για την ε, επιστήμη. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη. Ε, μπορεί να μας δώσει δυνατότητα να υπάρξει μεταφορά γνώσης. Ε, και επίσης ε, ε, τα χρήματα του φορολογούμενου θα μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει, στήριξε το παρελθόν όλα αυτά τα θέματα, αλλά ακόμα υπάρχει πολλής δρόμος πριν επιτύχουμε το στόχο της ανοιχτής επιστήμης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορεί να στηρίξει την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία έτσι ε, ώστε να συμπεριλαμβάνεται στις ε, προσπάθειές της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστώ την Επίτροπο. Θέλω να κάνω μία ανάλυση και μετά μία ερώτηση. συμβαίνει και ε, σε αυτά που λέει το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και σε άλλες αναλύσεις ότι τα κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία ε, δεν κατανέμονται ισόποσα. Ε, γεωγραφική η ανισορροπία ανάμεσα σε χώρες που οι μεν είναι πρωτοπόροι και οι άλλοι υπολείπονται. Υποτίθεται ότι υπάρχει κάποιο εργαλείο για να υπάρχει και πιο ε, ισότιμη κατανομή. Εμείς αυτό καταγράψαμε και ε, πράγματι υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια, κυρίως όσον αφορά ε, στην διαχείριση των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα γνωρίζει όλα αυτά και τι προτίθεται να κάνει για να αποφύγει τέτοιου είδους ανισορροπίες. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που είστε εδώ. Το Μάρτιο η νέα Επιτροπή θα δημοσιεύσει τη νέα στρατηγική για τη ΜΜΕ και ε, για την βιομηχανική τη στρατηγική. Και οι περάσινοι ζητούν αυτή η στρατηγική να στοχεύει μηδενικές εκπομπές και να μετατρέψει ε, την βιομηχανία, θεωρώντα ότι παίρνει περίπου 25 χρόνια να μετασχηματιστεί η βιομηχανία και θεωρώντας ότι κάποιε βιομηχανίε ε, του χάλιβα, των χημικών, είναι ενεργοβόρε βιομηχανίε και εκπέμπουν ε, μεγάλε ποσότητε εκπομπέ, μήπω η Κομισιόν ε, θα συμβάλλει στην απανθράκωση αυτών των βιομηχανιών και ποια μέσα θα υλοποιηθούν συγκεκριμένα θα προωθήσετε τα clusters του δεύτερου άξονα για να δώσετε προτεραιότητα και θα προσαρμόσετε το στρατηγικό ε, σχεδιασμό του ορίζοντα για να ε, υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την απανθράκωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και Επίτροπε. Όταν ε, μελετάμε το θέμα της βιομηχανίας και της ανταγωνιστικότητας, η εκπαίδευση και η καινοτομία είναι βασική σημασία. Χαίρομαι που έχουμε μία επίτροπο, έναν επίτροπο που είναι αρμόδιος για όλους αυτούς τους τομείς μαζί. Όταν μιλάμε για την έρευνα και την εκπαίδευση και την καινοτομία, βέβαια τα κράτη-μέλη έχουν την κυριότητα αρμόδιότητα. Βέβαια έχουμε το πρόγραμμα Ορίζοντα, στηρίζω όλους τους προλαλήσαντες ε, συναδέλφους που στήριξαν τις προτάσεις μας ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό κατά 50% τον προϋπολογισμό του ορίζοντα ε, για το 2021. Η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα κράτη-μέλη και τις μεταρρυθμίσεις μέσα από το εξάμεινο, όταν μιλάμε για θέματα εκπαίδευσης, καινοτομίας και έρευνας. Πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, αυτές τις συστάσεις, για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη με αυτόν τον τρόπο και μια άλλη ερώτηση σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί τώρα προετοιμάζεται και στρατηγική των ε, των μικρομεσαίων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, πώ θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τις παραδοσιακές ΜΜΕ θα μπορούσαν να υποφεληθούν τη ψηφιοποίηση, διότι είναι μεγάλο άλμα για αυτές. Ευχαριστώ, κύριος Ρομπέρος. Εγώ δεν θα μιλήσω για τα χρήματα, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο φάκελο αυτό σκιώδης. Έχω εργαστεί πάρα πολύ σκληρά και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια κομμάτια της διαδικασίας. Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να κάνουμε πιο αποτελεσματικά και φιλόδοξα τα ερευνητικά προγράμματα. Δαπανάμε χρόνο και χρήματα σε θέματα ανευσημασίας. Οπότε εμείς προσπαθούμε να πιέσουμε τις μικρομεσαίε επιχειρήσει να ακολουθούν διαδικασίες, ενώ θα έπρεπε να μας αφορούν τα παραδοτέα. Οπότε χρειαζόμαστε να δούμε τι χρειάζονται ε, για να τα πάνε καλύτερα οι επιχειρήσει αυτές. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Να επιμένουμε πως όλοι οι πόροι να είναι ευρωπαϊκοί. Όλα τα κεφάλαια, για παράδειγμα. Ακολουθήσαμε λοιπόν μια, μια διαδικασία όπου τα λιγότερα υποσχόμενα project από μια κατάλογο 20 ε, αφαιρέθηκαν και μετά δώσαμε επιδοτήσεις ανάλογα με τις επιδόσεις. Ε, αυτό είναι καλό γιατί έτσι μειώνουμε τη γραφειοκρατία και κάνουμε πιο επιχειρηματικές ε, επιλογές. Θα στηρίζατε κάτι τέτοιο. Έχετε το λόγο, συνάδελφε και όλοι μας εδώ ανησυχούμε για τις περικοπές που προτείνονται στον προϋπολογισμό, αλλά πείτε μου, καταρχήν η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το ποιο θα είναι η, ποια θα είναι η προτιμόμενη κατανομή των περικοπών. Υπάρχουν οποιαδήποτε ε, ε, θέματα τα οποία ε, να είναι απολύτως ασφαλή ε, να μην μπορεί να τα ακουμπήσει κανείς. Και μετά για την αναγόνηση του ευρωπαϊκού χώρου ε, έρευνας έχουμε και τις συνδεδεμένες χώρες εδώ ή μόνο τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Χρήστοφ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε επειδή ε, πρόκειται να επενδυθούν 300 ε, εκατομμύρια ευρώ στο ε, πρόγραμμα Horizon 2020, μιλάμε για πάνω από 60 πιλωτικά προγράμματα για την τεχνολογία 5G. Έχοντας αυτά κατά νου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προτείνει διάφορα προγράμματα για να ε, στηριχθεί αυτή η τεχνολογία της πέμπτης γενιάς τηλεπικοινωνιών, το 5G. Επίσης, ε, τώρα ήδη αρχίζουν να τρέχουν προγράμματα για την επόμενη γενιά, την έκτη γενιά, το 6G. Όμως θέλω να ρωτήσω, η επιπτώση στην υγεία από την τεχνολογία 5G οι επιπτώσεις δεν έχουν εξεταστεί και υπάρχουν ανησυχίες για το ε, πώς θα επηρεάσουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία της πέμπτης γενιάς στην ανθρώπινη υγεία. Έτσι λοιπόν ε, πρόκειται να χρηματοδοτήσετε προγράμματα όπου θα αναζητηθούν επιπτώσεις ε, στην υγεία. Ο κύριος Μπούζεκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι οι αποστολές μας. Σε ποια φάση προετοιμασίας βρισκόμαστε από επιστημονική και τεχνική άποψη. Αναφέρομαι σε πέντε. Βεβαίως, ε, η πρώτη σημαντικότερη αποστολή μας ε, είναι ε, το να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο. Δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά τις ε, περικοπές στον προπολογισμό. Όταν έχουμε σημαντικές ε, περικοπές, ε, αυξάνονται οι κίνδυνοι και οι χώρες όμως οι οποίες θέλουν κάποια διεύνηση των προγραμμάτων τους είναι αυτές οι οποίες έχουν άμεσα συνδεθεί με την Πράσινη Συμφωνία. Άρα περικοπές στη διεύρυνση και επιτείνεται ε, η τροτότητα ε, ορισμένων χωρών λόγω της πράσινης συμφωνίας. Πώς προτίθεστε να λύσετε το πρόβλημα. Η κυρία Επίτροπος ε, έχει το λόγο. Πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά. Αλλιώς μετά θα πρέπει να περάσουμε στα αγγλικά, εκτός αν οι μας δώσουν κάποια παράταση. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να πω ότι εκεί που δεν μπορώ να απαντήσω, εγώ και η ομάδα μου παραμένουμε στη διάθεσή σας για να παρέχουμε όσες πληροφορίες μπορούμε, διότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις ε, είναι σημαντικές γιατί έχουμε πραγματικές ανταλλαγές και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και η, ομάδα μου είναι στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις στο θέμα των αποστολών που είμαστε οι πέντε αποστολές έκαναν 24 συνεδριάσεις από το Σεπτέμβριο. Κάθε αποστολή είναι σε διαφορετικό στάδιο αλλά θα ε, υπάρξει μια κοινή συνάντηση μαζί μου όπου θα είμαι πολύ σαφής. Μέχρι τον Μάιο Κάθε αποστολή θα πρέπει να εντοπίσει την πρώτη δράση που θα πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε αυτή η δράση να μπορεί να συζητηθεί από το Κοινοβούλιο, από τους πολίτες και να μπορούμε να ε, δούμε, λαμβάνοντα υπόψη τα κριτήρια που έχει θέσει το Ευρωκοινοβούλιο και στη διαπραγμάτευση, ότι είμαστε σε θέση να έχουμε αποτελέσματα μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει. 2021-2024 αποτελέσματα που πρέπει να είναι ορατά για κάθε πολίτη, θα πρέπει να είναι καταμετρήσιμα κάθε χρόνο και έχουμε και τον περιορισμό του προπολογισμού 10% του ετήσιου. Από πλευρά μου, αυτό που είναι σημαντικό, ε, από τον Δεκέμβριο κάθε αποστολή έχει ορίσει ένα άτομο αρμόδιο για το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην διστάσετε να τους βρείτε. Ξέρουν ότι είναι εκεί για, για για το Κοινοβούλιο. Κάποιες αποστολές πρέπει να τονωθούν. Βέβαια, η αποστολή για ε, την καταπολέμηση του καρκίνου είναι ε, η πιο προχωρημένη. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον καθηγητή Ρικιάρτη, που είναι επικεφαλή ε, του Συμβουλίου, και έχουμε συζητήσει επί μακρόν την πραγματική ανάγκη να εντοπίσουμε δράσει συγκεκριμένε. Αλλά να μην ξεχάσουμε και από την αρχή να εμπλέξουμε και του πολίτε, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τι διαφορέ υποδομών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την πρόσβαση στι υπηρεσίε. Υπάρχουν ερωτήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και ε, είναι πολύ καλό να μιλάμε για επακριβία σε ιατρική, αλλά υπάρχουν ε, περιοχές του κόσμου ότι δεν υπάρχει ε, σύνδεση με το διαδίκτυο για να μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και θέματα, γι' αυτό σας καλώ να θέσετε κι εσείς αυτά τα ερωτήματα και τον Μάιο θα δούμε τις πρώτες αντιδράσεις για να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα εις βάθος τη συζήτηση. Ε, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα, η κυρία Μιχαήλοβα μου θέσατε το ερώτημα, αλλά και ο κύριος Μπούζεκ για τα widening measures, τα διευρυντικά μέτρα. Δεν υπάρχει ε, κάτι το οποίο... Ε, αυτό το, το θέμα διεύρυνσης είναι μεγάλη προτερότητα, διότι είναι σημαντικό. Ε, οι αριθμοί είναι εκεί. Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην καινοτομία και την έρευνα στο θέμα του προγράμματος του ορίζοντα 900 εκατομμύρια ευρώ για τις χώρες διεύρυνσης. Έχουμε 5,6% του ορίζοντα για τα EU13, το υπόλοιπο για τους 15. Τώρα, χάρη στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε τη δυνατότητα να τα αλλάξουμε. Και γι' αυτό περισσότερα μέτρα έχουμε. Ε, θα συνεχίσουμε αυτά που δουλεύουν και έχουν αποτέλεσμα. Το teaming, το twimming, το cost κλπ. Εδώ με απασχολεί να δούμε πώς να διασφαλίσουμε τη συνέργεια με το ε, ΕΤΠΑ έτσι ώστε να υπάρχει μια διαφορετική δυναμική. Διότι είναι ε, ωραίο να εξηγούμε στις περιφέρειες ότι θέλουμε να έχουμε κέντρα υπεροχής και αριστείας, αλλά πρέπει να υπάρχει το κτίριο, το εργαστήριο, να είναι εξοπλισμένα, να δουλεύουν στις συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να προωθήσουν τις ιδέες τους και έτσι ώστε αυτές οι ιδέες να μετατραπούν σε προϊόντα. Θα ήθελα να προτείνω δύο άλλα ε, μέσα. Την προεπαλήθευση των έργων. Ορισμένα έργα χρειάζονται λίγο ε, για να ε, προτού απορριφθούν στη χρηματοδότηση και θα ήταν καλό να υπάρχει ένας μηχανισμός για να ενταχθούν υπάρχοντα κονσόρτσια και συμπράξεις. Είναι πολύ περίπλοκο. Υπάρχουν ε, κονσόρτσια που ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί ο ορίζοντας. Ε, θα πρέπει ε, η πρόθεσή μου είναι να δώσουμε κίνητρα και από τις δύο πλευρές για να ανταλλάξουμε πραγματογνωμοσύνη, να υπάρχουν συνέργειες και να κάνουμε κοινά προγράμματα. Και είναι κάτι το οποίο θέλω να συνεχίσω να προωθώ. Επίσης, θα ήθελα να αναστοχαστούμε εδώ και να μην ξεχνάμε την ε, πλευρά της εκπαίδευσης. Οι δράσεις Marie Curie. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ανάμεσα στις δύο γενικές διευθύνσεις, ΕΑΚ και RNI, που μας επιτρέπει να χρηματοδοτούμε ερευνητές που δεν κατόρθωσαν να πάρουν χρηματοδότηση στον ορίζοντα 2020, μπορούμε να έχουν μια υποτροφία έτσι ώστε να κάνουν την έρευνά τους σε μία από τις χώρες της ΕΕ13 και ιδιαίτερα στη χώρα προέλευσής τους. Έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, εκπληκτικά. Έχουμε χώρες όπου η απόδοση αυτών των ερευνητών είναι πάνω από το 70% και με βέβαιη ότι στο τέλος αυτής της διετίας ε, της πιλωτικής θα τους αξιολογήσουμε και θα έχουμε μια βάση για να κτίσουμε ένα μηχανισμό που θα είναι μόνιμος. Ε, πιστεύω ότι θα ήθελα να συνεχίσω να ε, δουλεύω προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω και για το Συμβούλιο ε, των, το Ευρωπαϊκό των Καινοτομιών και των ΜΜΕ. Θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να είναι ενημερωμένες όσο δυνατόν περισσότερο και εδώ στρέφω τον, την, το, το βλέμμα στο OIT. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας δουλεύει καλύτερα με το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό για την Καινοτομία. Η πρώτη αποστολή του OIT είναι να κτίσει οικοσυστήματα. Θα το ξανασυζητήσουμε εδώ αυτό και θα δούμε διαφορετικέ και διστάμενε απόψει. Αλλά να πάει και σε αυτού να εντοπίσουν του πρωταθλητέ, του μελλοντικού ε, ε, πρωταθλήτες έτσι ώστε να περάσουν πιο εύκολα στο ε, Συμβούλιο και να ζήτησα από την ομάδα μου να δουλέψουμε έτσι να δούμε πώς να φτιάξουμε γέφυρες ανάμεσα στο έργο του OIT και το έργο του OIC. Και εδώ ευστώ την προσοχή σε ένα θέμα που δεν ακούσαμε, το θέμα των γυναικών καινοτόμων. Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου δείχνουν ότι τα προγράμματα στα οποία υπάρχουν γυναίκες είναι 7-8%. Είναι απαράδεκτος αυτός ο αριθμός. Ζήτησα από τις ομάδες μου, από τώρα και στο εξή, να έχουμε ένα στόχο 20%. Να υπάρχουν ε, στις ε, συνεντεύξεις τουλάχιστον γυναίκες καινοτόμοι, γυναίκες ε, διευθύντρες επιχειρήσεων που να μπορούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Και θα αποφασίσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την απόφαση στην επόμενη πρόσκληση. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Θα ήθελα άλλη μια φορά να σας πω πόσο αναγκαίο είναι να στηριχτώ σε εσά του επόμενου μήνε για να έχουμε μια πραγματική ε, περισυλλογή και μελέτη στο νέο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Γιατί? Γιατί έχουμε τους τρεις πυλώνες του ορίζοντα. Αυτοί οι τρεις πυλώνες θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους επιτέλους. Βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και το Μαρκιουρί μπορούν να μας βοηθήσουν πώς να δούμε θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια ανάμεσα σε όλους. Πώς η IT και το European Innovation Council θα μπορεί να μας επιτρέψει να έχουμε ε, τους στόχους μας. Είναι πολύ καλή φιλοδοξία, αλλά δεν θα επιτευχθεί. Οι αποστολές και πάλι δεν είναι οντότητες ε, ξεχωριστές, απομονωμένες. Έχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα κονδύλια και με άλλα ταμεία και με τις ε, και συνεταιρισμούς. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε την ευκαιρία με την απλούσευση, με περισσότερη σαφήνεια να προχωρήσουμε. Και στο πλαίσιο όλων αυτών ε, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τους τρεις πυλώνες με τις συνέργειες, αλλά από κάτω έχουμε το τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Παιδείας. Ε, είναι πολύ καλό να μιλάμε για το πόσο λείπουν οι δεξιότητε, αλλά στη βάση έχουμε τα συστήματα τα εκπαιδευτικά. Γι' αυτό πρότεινα ότι η μέρα καινοτομία και έρευνας να περιλαμβάνει ένα κοινό πάνελ για να δούμε τις συνέργειες. Ε, θα έχουμε και επίσης ε, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο θα δημοσιευτούν οι στόχοι του European Research Area και του European innovation area. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι σαφεί συνέργειε, όπως είπε η κυρία Σπυράκη, για τα παιδιά, για την προστασία, για το ρόλο των γονιών, των οικογενών. Αυτό είναι ένα σχέδιο δράσης ψηφοποίηση. Θα πραγματοθεί τον Ιούνιο. Ανήκει και σε θέματα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και ε, στο χώρο της εκπαίδευσης. Σας καλώ τους επόμενους μήνες λοιπόν να ε, θέλετε ε, τα ερωτήματά σας, να είστε επικριτικοί και να συνεχίσουμε επικοδομητικά έτσι ώστε αυτό το πρώτο χρόνο με όλους τους περιορισμούς που έχουμε αλλά χωρίς να δεχτούμε άλλες περικοπές στον προπολογισμό, να θέσουμε σταθερές βάσεις, έτσι ώστε να προχωρήσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ για τον εξαιρετικό διάλογο. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υλοποίηση του ορίζοντα και να συνεργαστούμε ε, στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.